Okay, if, if the uh, photographers could take a discreet distance too, that would be appreciated. Και αν παρακαλώ μπορούσαν οι φωτογράφοι να απομακρυνθούν λιγάκι, πολύ θα το εκτιμούσα και θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση λοιπόν τώρα. Καταρχάς θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται ούτω η ημερήσια διάταξη. Πρωτού προχωρήσουμε στις κυρίως εργασίες μας. Yeah. Έχω μία ανακοίνωση λυπηρή να σας κάνω, να σας ενημερώσω όλους τους παράγοντες σήμερα το πρωί. Ο Μίγκουελ Πόρτας, της ομάδας της ΓΚΟΕ, μέλος της Επιτροπής μας, ο οποίος ήταν ενεργό στην Επιτροπή μα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα νομισματικού διαλόγου και ο οποίο ήταν επίση συντονιστή στην Επιτροπή προπολογισμών, απεβίωσε χθε. στην ηλικία των μόλις 53 ετών. Και στη μνήμη του σας ζητώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Um, Στη συνέχεια, έχω κάποιες άλλες σύντομες ανακοινώσεις, όπως τα γνωρίζετε. Θέλαμε να ψηφίσουμε διάφορα σχέδια εκθέσεων σήμερα το απόγευμα, αλλά αναβλήθηκε για την επόμενη συνάντηση και για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί η γραμματεία σας έχει διανέμει ε, το νέο σχέδιο ημερήσιας διάταξης με τις αλλαγές. Αύριο το απόγευμα λοιπόν θα έχουμε πιο σύντομη ημερήσια διάταξη λόγω των αλλαγών αυτών που έλαβαν χώρα. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 9 η Ιανουαρίου, 16 Ιανουαρίου, 6ης Φεβρουαρίου, 12 η Μαρτίου. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, τις έχουμε, τα έχουμε διανύμει τα πρακτικά, θεωρώ ότι έχουν εγκριθεί. Σας ευχαριστώ και τώρα θα περάσουμε στον ε, διάλογο των νομισματικών θεμάτων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και χαίρομαι ιδιαιτέρω που καλωσορίζω τον Μάριο Ντράγκη στην Επιτροπή μα, Ο προηγούμενο διάλογο των νομισματικών θεμάτων ήταν στι 19 Δεκεμβρίου. Τελευταία συνεδρίαση και η επόμενη συνεδρίαση είναι η 9η, θα γίνει στις 9 Ιουλίου. αν Ανυπομονούμε λοιπόν ήδη και όπως ξέρετε θα μας μιλήσει πρώτα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ειδικής Τράπεζας και μετά θα ακολουθήσει η συνήθις ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι το λέγω έχει ο Μάριο. Thank you. Madam Chair, members of the Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ πάλι στο Κοινοβούλιο μπροστά από την Επιτροπή σας για την ε, τακτική ανταλλαγή απόψεων. Σύμφωνα με την ε, αλλαγή της κατάστασης πρέπει να σας πω ότι υπάρχει υπάρξει αύξηση 430 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η Ευρωζώνη έχει διαπράξει, α, το, έχει διαλέξει το ρόλο της έχοντας χορηγήσει 150 εκατομμύρια ευρώ πλένο Χαίρομαι που τώρα οι υπόλοιποι ε, μετόχοι έχουν προσφερθεί να συμμετάσχουν και αυτοί ε, στην αύξηση των πόρων. Είναι λοιπόν πρωταρχική σημασία ο μηχανισμός ευρωπαϊκής σταθερότητας να γίνει απόλυτα λειτουργικός. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να υποστηρίξει το μηχανισμό αυτό. Βεβαίως, ακόμη και με μέτρα προστασίας πολύ σημαντικά τα οποία θα θέσουμε σε λειτουργία, οι χώρες της Ευρωζώνης πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν διαρθρωτικές και ε, χρηματοπιστωτικές προσαρμογές που είναι απαραίτητες. Ως συνήθως ε, αρχικά θα επισέλθω στην ε, τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Στη συνέχεια θα αφιερωθώ στα θέματα τα οποία ε, προτείνετε εσείς οι ίδιοι. Εκτίμηση και αξιολόγηση των ειδικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και αξιολόγηση των οικονομικών ε, καταστάσεων στην ε, νομισματική ένωση. let me first focus on και θα ήθελα καταρχάς να κοιτάξουμε τις ε, οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη από την τελευταία μας συνάντηση στις 19 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Οι δείκτες που είχαμε στη διάθεσή μας για το πρώτο τρίμηνο του 2012 επιβεβαιώνουν την σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας σε χαμηλά ωστόσο επίπεδα. Οι πρόσφατες εξελίξεις στα δεδομένα που προκύπτουν από τις έρευνες είναι ανάμεικτα και τονίζουν ότι υπάρχει αστάθεια και βεβαιότητα. Όσο για το μέλλον, η ανάπτυξη θα πρέπει να υποστηριχθεί από την εξωτερική ζήτηση, από την αλλοδαπή ε, ζήτηση, από πολύ χαμηλά επιτόκια και από έκτακτα μέτρα εκ παραλίλου, κίνδυνοι περαιτέρω ύφεσης, προκύπτουν ιδιαίτερως από μία ανανεωμένη εντατικοποίηση των εντάσεων στην ε, αγορά των εθνικών αγορών και ενδεχόμενες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, ενδεχόμενες ε, μελλοντικές περαιτέρω αυξήσει των τιμών των βασικών προϊόντων, επίσης μπορεί να παρεμποδίσουν την οικονομική δραστηριότητα. Ε, ο πληθωρισμός ήταν 2,7 το Μάρτιο στην Ευρωζώνη, ε, απαράλλακτο σε σχέση με τους τρεις προηγούμενους μήνες και ο πληθωρισμός ε, ενδεχομένως κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει πάνω από 2% κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους λόγω των αυξήσεων των τιμών ενέργειας και των έμεσων φόρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθεί να αναμένει ετήσια επιτόκια κάτω από το 2% για τις αρχές του 2013 σε ό,τι αφορά το μέλλον, σε ένα περιβάλλον ε, περιορισμένης ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και συγκεκριμένων ε, ε, αναμενόμενων εξέλιξεων σε ό,τι αφορά την, τον πληθωρισμό, οι τιμές θα υποστούν πιέσεις. Μέτριες, ωστόσο. ενδεχόμενοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από τις ε, τιμές του πετρελαίου και από άλλες ε, αυξήσεις των, ε, των φόρων. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα δείξει ιδιαίτερη προσοχή σε οποιοδήποτε ενδείξει μεταβίβαση των τιμών, των υψηλών τιμών της ενέργειας, στους μισθούς, στα κέρδη και γενικά στην καθοτρισμό των τιμών. Και είναι απαραίτητο σε ό,τι αφορά τι μεσοπρόθεσμες ε, προσδοκίες για τον πληθωρισμό να παραμείνουν ε, βασικά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Η νομισματική ανάλυση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, ανάπτυξη της ζήτησης του χρήματος, επιβεβαιώνει τις εξελίξεις των τιμών που θα παραμείνουν στα πλαίσια τη σταθερότητα των τιμών. Τα δεδομένα για τα χρήματα και για τις πιστώσεις μέχρι το Φεβρουάριο υποδεικνύουν μια σταθεροποίηση των ε, οικονομικών όρων και παράλληλα η ζήτηση για πιστώσεις παραμένει αδύναμη λόγω της περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας και της συνεχιζόμενης ε, διαδικασίας προσαρμογής των εσολογισμών στους μη ε, χρηματοπιστωτικούς κλάδους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι τράπεζες να ενισχύσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητά τους, διαπτυρώντας και ε, μάλλον ε, παρακρατώντας μπόνους. Γιατί το πόσο σταθερά θα είναι τα έγγραφα ισολογισμού των τραπεζών θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την ε, πίστοση στην οικονομία και στον ε, εξορθολογισμό της χρηματοδότησης. Και τώρα θα ήθελα να στραφώ σε θέματα αποτελεσματικότητας το τελευταίο, των τελευταίων μέτρων, ε, εκτάκτων μέτρων νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος σε ό,τι αφορά τις ε, LTROs, τις μακροπρόθεσμες ε, δράσεις επαναχρηματοδότησης. Θα ήθελα καταρχάς να είμαι σαφής γιατί εφαρμόσαμε τις λειτουργίες αυτές σε τριετή βάση. Όπως θα θυμάστε, το δεύτερο ήμιση του 2011 ε, χαρακτηρίστηκε από μια εντατικοποίηση της έντασης σε ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες ε, αγορές και το δημόσιο χρέος και ένα περιβάλλον υψηλής ανασφάλειας. Αυτό παρεμπόδισε την πρόσβαση στις τράπεζες, των τραπεζών της Ευρωζώνης σε χρηματοδότηση. Αν δεν είχε ληφθεί δράση, αυτό θα μπορούσε να είχε αποτέλεσμα ε, μεγάλες Και στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Τα LTRO απάλυναν κάπως αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, αυτές οι πράξεις ε, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης οι τράπεζες κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις επικρόστατες ανάγκες ρευστότητας που εκτιμούνται περίπου σε 520 δισεκατομμύρια αφαιρώντας ρευστότητα από άλλες δραστηριότητες. Επίσης, οι τράπεζες επωφελήθηκαν από την αυξανόμενη ασφάλεια σε ό,τι αφορά την μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση χάρη στην ε, ε, μεγαλύτερη διάρκεια των νέων επιχειρήσεων. Καταλαβαίνω ότι είστε ιδιαίτερα ενδιαφέρον σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μεταβίβαση και η επίπτωση των πράξεων μακροπροθεσμής χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία. Και όντως είναι κρίσιμο το σημείο αυτό. Η διασφάλιση ότι η πολιτική η νομισματική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξακολουθεί να μεταφέρεται με αποτελεσματικό τρόπο στην, στην πραγματική οικονομία ήταν ένας παράγοντας κλειδί σε ό,τι αφορά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και είναι ενθαρρυντικό ότι βλέπουμε ότι μεγάλο αριθμό μικρών τραπεζών συμμετείχαν σε αυτέ τι δύο πράξει. Οι μικρέ τράπεζε είναι σε καλύτερη θέση να επαναχρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα τι μικρομεσαίες επιχειρήσει που αποτελούν το μεγαλύτερο μοχλό ε, σε ό,τι αφορά και τις θέσει εργασία στην οικονομία. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι πλέον ότι η ρευστότητα τη Κεντρικής τράπεζα έχει προσεγγίσει πολύ την πραγματική οικονομία. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό από μόνο του θα δώσει όθηση στις, ε, στη δανειοδότηση των ε, επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Καταρχάς, η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να παρέμβει σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της ρευστότητα των τραπεζών, γιατί είναι δικό του ε, το θέμα. Αλλά θεωρούμε ότι θα επαναχρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, γιατί αυτό είναι ο ρόλο του τραπεζικού συστήματο. Κατά δεύτερον, η μεροδική εξέλιξη τη ανάπτυξη των πιστώσεων θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τη ζήτηση του τρέχον περιβάλλον, η ζήτηση κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει χαμηλή. Ω εκ τούτου, η ανάπτυξη και του χρήματο αλλά και των πιστώσεων μπορεί να παραμείνει ασθενή για κάποιο καιρό προτού βελτιωθεί η συνολική οικονομική κατάσταση. Και η μελέτη τη Τράπεζα για τη Δανειοδότηση με κάποια καινούργια στοιχεία θα δημοσιευθεί στι 10 σήμερα το πρωί. Κάποιοι εξημών ενδεχομένω να ανησυχείτε για τους ε, κινδύνους του πληθωρισμού προκύπτουν από αυτά τα έκτακτα μέτρα. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα δεν αποτελούν ε, περιορισμό σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Ειδικά να μην ξεχνάμε ότι τα επιτόκια για τα τριετή Τη πράξεις πράξη μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης δεν είναι καθορισμένα, αλλά συνδέονται με το βασικό επιτοκίο πολιτικής επιπλέον για να μετρήσουμε την νομισματική ρευστότητα δεν κοιτάμε ε, τον ισολογισμό του συστήματος, αλλά τον ισολογισμό του ίδιου τραπεζικού συστήματος, γιατί μόνο αυτό καταδεικνύει την σχέση με την πραγματική οικονομία και αυτό αποτυπώνεται από τα νομισματικά στοιχεία και από τα πιστοτικά στοιχεία, τα οποία, όπως ε, ανέφερα, εξακολουθούν να παραμένουν σε ύφεση. Να είστε σίγουροι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέτρα που έχει στην διάθεσή της για να καταπολεμήσει ενδεχομένου κινδύνους σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των τιμών σε περίπτωση που εμφανιστούν. Επίση ακούμε ανησυχίε ότι το ευρωσύστημα ε, ε, έχει εκτεθεί σε ε, εξαιρετικά μεγάλους κινδύνους και θα ήθελα να τονίσω ότι η επέκταση του ισολογισμού μας γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη σοφροσύνη και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε να αναφερούμε την πρόσθετη μας ε, νομιμότητα και το πλαίσιό μας. Επιπλέον, η εφαρμογή μέτρων ελέγχου του κινδύνου, όπως τα κουρέματα σε όλα τα νομισματικά πολιτικά συστήματα, προστατεύει την ε, σταθερότητα των, της χρηματοοικονομικής θέσης μας. Θα ήθελα να σας πω επίσης κλείνοντας ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι έκτατα και προσωρινά και επιπλέον η υποστήριξη της ρευστότητας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις σωστές νομισματικές και διασχετικές πολιτικές για το κεφάλαιο που προκύπτουν από την ε, σταθερή ανάπτυξη και σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και τώρα θα ήθελα να περάσω στο τέταρτο θέμα να συζητήσω, αν θέλετε, τις μακροοικονομικές αστάθειες στην ευρωπαϊκή ε, ε, ε ζώνη. Φυσικά, η οι ανισορροπίες σε μια νομισματική ένωση και οι αποκλήσει είναι φυσιολογικέ. Παρατηρούνται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να γίνουν μόνιμες και να αποτελούν κομμάτι της γενικότερης δομής. Δυστυχώς, πολύ μεγάλες ε, ανισοσκέλειες επιτράπηκε να συσσωρευτούν τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτέ οι ανισοσκέλειες προήλθαν από διάφορες πηγές, ανεπάρκη δημοσιονομική πειθαρχία, χρηματοοικονομικέ ε, υπερβολές, ε, μη υλοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων, ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά στι αγορές εργασία και προϊόντων και σημαντικέ απώλειες ανταγωνιστικότητα. Όλες αυτά απαιτούν επίγουσα και αποφασιστική προσαρμογή είναι σαφώς ότι δεν μπορεί να είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, η αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών. Όσον αφορά την νομισματική πολιτική, στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη, στο συνόλο της για αυτό το σκόπο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί διαρκώς όλες τις σχετικές πληροφορίες από τις χώρες και τις διάφορες επιχειρήσεις της Ευρωζώνης. Ωστόσο, η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να εστιαστεί σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αποκλήσεων μεταξύ μεμονωμένων χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό είναι το καθήκον κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να προβούν σε αποφασιστικές δράσεις πολιτικής για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αδυναμίες στους δημοσιονομικούς, χρηματοπιστωτικούς και διαρθρωτικούς τομείς. Σημειώνουμε ότι σημειώνεται πρόοδος σε πολλές χώρες. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να συμπληρωθούν σήμερα με μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές οι οποίες θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και θα, θα διευκολύνουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, τις νεοσυσταθήσεις επιχειρήσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και εδώ οι κυβερνήσεις θα πρέπει να γίνουν πιο φιλόδοξες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ε, για την ενίσχυση του, οικονομικού, του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Έχουν ενισχυθεί οι δημοσιονομικοί κανόνες στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η εισαγωγή του Δημοσιονομικού Συμφώνου για το οποίο μιλήσαμε στο Κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο και υλοποιούμε τη νέα εστίαση διόρθωση των μακροοικονομικών ανισοσκελιών. Η πρόσφατη κρίση έχει δείξει ότι μία ε, νομισματική ένωση που λειτουργεί σωστά δεν χρειάζεται απλά ισχυρή θεσμική βάση με την νομισματική πολιτική στο κέντρο, αλλά και ε, μια ισχυρή βάση για τις οικονομικές πολιτικές. Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης πρέπει να θεωρείται κοινή ευθύνη. Είμαι βέβαιος ε, ότι πολλοί από εσά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσετε ότι χρειαζόμαστε αλλαγή νοοτροπίας όταν χαράσουμε και διεξάγουμε πολιτική. Και στον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε. Οι οικονομικές πολιτικές ε, της Ευρωζώνης ε, είναι εν τέλει εγχώρες πολιτικές της Ευρωζώνης ακριβώς λόγω των, ε, πιθανότητων διάδοση θα πρέπει να παρακολουθούνται διαρκώς και να διορθώνονται για το συλλογικό συμφέρον της Ευρωζώνης. Αυτό θα πρέπει να ισχύει τόσο στι δημοσιονομικέ όσο και στι μακροοικονομικέ πολιτικέ. Αλλά η επιτήρηση από μόνη τη δεν επαρκεί. Οι πολίτες αναμένουν επίσης από την Ευρώπη κοινέ απαντήσει για τις κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης. Σε ένα πλαίσιο παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκού δημοσιονομική εξυγίανση, οι χώρες της Ευρωζώνης θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Δεδομένου ότι έχουν ένα κοινό νόμισμα, έχουν ακόμα περισσότερου λόγου από άλλε χώρε να συνεργαστούν. Αυτή η συνεργασία μπορεί να γίνει στην έρευνα, την ανάπτυξη, την παιδεία ή την υποδομή. Θα πρέπει να αγωνιστούν για τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία. Επιτρέψτε να προσθέσω ότι ακριβώς όπως και στην περίπτωση της ανταγωνιστικότητας θεωρώ ότι και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί κοινή ευθύνη σε μια νομισματική ένωση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης παρατηρήσαμε αρνητικές ε, περιπτώσεις διάδοσης στις διάφορες χώρες της Ευρωζώνης ε, και μεταξύ των ε, τραπεζικών τομέων, του τραπεζικού τομέα και των αντίστοιχων δημοσίων χρεών. Οι εθνικές επόπτικες αρχές αντιμετώπισαν το γνωστό πρόβλημα ότι στους, σε καλούς καιρούς οι μεγάλες τράπεζες λειτουργούν ως ευρωπαϊκοί θεσμοί και σε κακούς καιρούς ε, κατηγορούνται. Η διασφάλιση μιας νομισματικής ένωσης που λειτουργεί καλά συνεπάγεται ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών και αποφασιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει φέρει ειρήνη και ευημερία, ενώ μου είναι δύσκολο να ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης την οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να οριστεί. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε ακόμη περισσότερα για την μακροπρόθεσμο όμως όραμα για την Ευρώπη όπως κάναμε στο παρελθόν σε άλλες καθοριστικές στιγμές της ιστορίας της Ένωσής μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Μάριο και τώρα θα περάσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις με τη γνωστή διαδικασία. Τα ρακαλώ τα μέλη να διατηρούν τις ερωτήσεις τους σε όχι περισσότερο από 1,5 λεπτό και Μαρίο θα χρειαστεί να απαντήσετε εντός 3,5 λεπτών δηλαδή σε κάθε ερώτηση ώστε να έχουμε ε, τμήματα 5 λεπτά ουσιαστικά. Θα ξεκινήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ε, ε Επιτροπής εκ μέρους του ΣΕΛΚ, τον Πάμπλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ντραγιόλη. Συμφωνούμε σχεδόν ότι για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση θα πρέπει να βελτιώσουμε τα δημοσιονομικά μας, να εξηγιάνουμε τα δημοσιονομικά μας και αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Ε, ένα από τα προγράμματα, τα κυρίες χώρες που έχει πρόβλημα είναι η Ισπανία, αλλά είναι, έχει αναλάβει σοβαρές δεσμεύσεις για την δημοσιακή δημοσιονομική της εξυγίανση με πολλά μέτρα. Ποτέ σε μια χώρα δεν είχαν καταβληθεί τόσες μεγάλες προσπάθειες μεταρρύθμιση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να αλλάξουν τα πράγματα. Αναμφίβολα κυρία Ντράγκε, αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όντως θα πρέπει ε, να αναγνωριστεί η προσπάθεια αυτή και να αποδείξετε πόσο μπορείτε να μας υποστηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια. Και βεβαίως ε, η Ισπανία δεν είναι η χώρα που ελέγχει πλήρως το όλο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει πολύ περισσότερα πράγματα. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα έχει ε, φαντάζομαι ότι θα έχει κάποιες ε, επιπτώσεις ε, στην ανάπτυξη, αρνητικές. Αλλά θα έχουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μεγάλα ωφέλη. Αναμφίβολα όλες οι προσπάθειες θα καταλήξουν σε αποτελέσματα και θα μπορέσουμε και πάλι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνεχίσουν όλες οι χώρες που έχουν τα συστήματα να καταβάλουν προσπάθειες. Σε αυτές τις χώρες βλέπουμε ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι καταβάλουν προσπάθειες και πρέπει να ε, συνεχίσουν να τις καταβάλουν. Εσείς από τη μεριά σας κύριε Ντράγκη τι θα κάνετε, θα ενεργήσετε, θα μπορέσετε να παρέμβετε στις δευτερογενείς ε, αγορές χρέους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχή ότι συμφωνώ απολύτω μαζί σας. Οι προσπάθειες που καταβάλει αυτή τη στιγμή η Ισπανική κυβέρνηση, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, δεν μπορούμε αν συνεχίζονται οι ιδιωτικές συζητήσεις να κάνουμε σοβαρή κουβέντα εδώ. Παρακαλώ. Διερωτώ κι εγώ. Τι συνέβη ξαφνικά, λέει ο κ. Δράγκη. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και με αυτά τα οποία είπατε στην αρχή της παρέμβασής σας. Η κυβέρνηση της Ισπανίας όντως καταβάλει, όπως είπατε και εσείς, εξαιρετικές προσπάθειες και έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο και βεβαίως συνεχίζονται αυτές οι προσπάθειες και τώρα είναι συνεχόμενες προσπάθειες και δεν έχουμε λόγους να αμφιβάλλουμε για την πλήρη δέσμευση της Ισπανικής κυβέρνησης ότι θα θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Κατά την άποψή μου όλοι είναι κοντά στην Ισπανία σε αυτό το εγχείρημα. θα έχω την δυνατότητα να σας εξηγήσω πώς έχουν αυτές οι LTROs, οι πράξεις για πιο, πιο μακροχρόνιας χρηματοδότησης. Όπως ξέρετε, τα δικά μας τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά για αρκετό ε, χρονικό διάστημα. Εσείς μιλήσατε ενδεχομένως για επαναδραστηριοποίηση του LRP. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι εμείς βασικά πρέπει να ενεργούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μας δίδει η συνθήκη και η δική μας εντολή είναι να δούμε κατά πόσον επιτυγχάνεται και με και η σταθερότητα των αγορών. Όπω καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι αντικείμενο πολύ ευάλωτων ισορροπιών. Θέλουμε εμείς να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για το λόγο αυτό πρέπει να ενεργούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Δεν θα είναι καλό ούτε για μας, αλλά ακόμη περισσότερο για την αξιοπιστία μας και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσουμε τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μας δίδει η συνθήκη και να ξεπεράσουμε την εντολή. Ευχαριστώ τώρα για την ομάδα των σοσιαλιστών να σας άλλος ο αντιπρόεδρος, η κυρία Μακάρθη. Ευχαριστώ. Θα συμφωνείτε, Πρόεδρε, ότι η κρίση είναι πλέον πολιτική βλέποντας την κατάρρευση της Ολλανδικής ε, κυβέρνησης. Πιστεύω ότι η ε, στις γαλλικές, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας γαλλικές εκλογές ε, μπορεί να θεωρηθεί κατηγορία της, του προγράμματος λιτότητας. Έχετε απορρίψει τις εκκλήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης. Θεωρείτε ότι έχετε βασιστεί υπερβολικά στα τριετή δάνεια Μήπως είναι ώρα να αλλάξετε πορεία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Thank you. Thank you. No, we don't believe. Ευχαριστώ. Όχι, δεν πιστεύουμε ότι η νομισματική πολιτική είναι υπερβολικά περιορισμένη. Θεωρούμε ότι είναι αρκετά ικανοποιητική Από ό,τι μαθαίνουμε από τις τραπεζικές μας έρευνες, ε, όσον αφορά τους περιορισμούς στην παροχή πιστώσεων από το τραπεζικό σύστημα, αυτοί έχουν μειωθεί σημαντικά από το περασμένο LTRO μέχρι σήμερα. Οι περιορισμοί λοιπόν αυτοί που αφορούσαν τα χρήματα που μπαίνουν στην οικονομία για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι αποκλειστικά, προέρχονται κυρίως από τη ζήτηση. Η ζήτηση για πιστώσεις. Ε, σε επαρκή χρόνο τα χρήματα αυτά θα βρουν το δρόμο τους προς την οικονομία για να τονώσουν, για να επαναδρομολογήσουν την ανάπτυξη και ο πληθωρισμός επίσης περιμένει περιορισμένος αυτή τη στιγμή. Η νομισματική μας πολιτική λοιπόν παραμένει ως έχει παρακολουθούμε ωστόσο όλες τις εξελίξεις και αποφασίζουμε ανάλογα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα για το ή Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνειδητοποιούμε ότι δεν σας είδαμε εδώ και κάποιο χρόνο, διότι η κατάσταση σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από τα Χριστούγεννα άλλαξε αρκετά. Δεν θέλω να κάνω επικρίσεις, απλώς θα ήθελα να σας πω το εξής. Γενικά πριν από τα Χριστούγεννα εμείς υιοθετήσαμε το περίφημο Six Packs λανσάρατε αυτό το LTRO, πράξεις για πιο μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, άλλαξαν τα πράγματα και υπάρχουν σήμερα κυρίως δύο θέματα που με απασχολούν και μιλώ εξ ονόματος και άλλων συναδέλφων. κρατημέλη βλέπουμε ότι δεν μπορούν να σεβαστούν τους στόχους. Εγώ στο Six Pack είχα μιλήσει πάρα πολύ για πειθαρχία, δεδομένου ότι πρόκειται για μια πραγματικότητα η οποία πλήττει χώρες όπως την Ολλανδία, που ήτανε ε, οι πρώτες στην καταπολέμηση των προβλημάτων που υπάρχουν. Δεύτερον, αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι βλέπω ότι μία από τις επιπτώσεις του LTRO, ίσως δεν το θέλαμε αυτό, είναι ότι οι τράπεζες τείνουν να αγοράσουν κρατικό χρέος. Και ο καθένας αγοράζει το δημόσιο χρέος του, κάτι το οποίο είναι όχι μόνο αντίθετο με αυτό που θέλουμε να κάνουμε στα πλαίσια ενιαία εσωτερική αγορά εδώ και χρόνια, αλλά όπω υπογράμισε και ο Τζόρτζο Σόρο, θα μπορούσε να έχει καταστροφικέ επιπτώσει την ημέρα που θα υπάρχει λιγότερη πραγματική αλληλεγγύη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Συγκεκριμένα λοιπόν σήμερα, χωρίς να πω ότι είναι εύκολο να ευρεθεί η κατάλληλη λύση, πώς αυτές οι δύο εξελίξεις που είναι ανισχυτικές κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να διορθωθούν. Έχουμε τα διάφορα κείμενα τα οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Ε, πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ξεφύγουμε από αυτά τα προβλήματα. Well, thank you, Σας ευχαριστώ. Μου κάνετε πραγματικά δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την λιτότητα. Αλλά ας κάνουμε μια άλλη ερώτηση. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα μπορούσε να αποφευχθεί. Πώς ήταν η κατάσταση στις αγορές και για ποιο λόγο άρχισε αυτή η δημοσιονομική εξυγίαση. Βασικά διότι αποφάσισαν οι αγορές ότι δεν θα χρηματοδοτήσουν το δημόσιο, το κρατικό χρέος. Διότι κατάλαβαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ε, ε, δεν μπορούσε να συνάδει με την αναλογία που είχε στο ΑΕΠ κάθε χώρα. Άρα ήταν κάτι το, το αναπόφευκτο ως μέτρο για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών. Το να αρνηθούμε τώρα ότι η δημοσιονομική εξυγίανση έχει κάποιες επιπτώσεις περιοριστικές και αρνητικές βραχυπρόθεσμα δεν είναι πραγματικότητα. Εάν λοιπόν έχετε τέτοιου είδους ε, επιπτώσεις στέρησης από τις αγορές, κατά κάποιο στέρησης από τις αγορές, ε? ας δούμε ε, την... ανεργία των νέων. Δεν είναι άμεση επίπτωση, δεδομένου ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο πιο μακροπρόθεσμα πλήττει τι αγορέ μα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Συγχρόνως να εφαρμόσουμε δομικές και διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές. Και δεν μιλούμε τώρα για οικονομίες οι οποίες πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν ανταγωνιστικές. Κάποιες χώρες από αυτές έχασαν την ενεργητικότητά τους και την ανταγωνιστικότητά τους. Το παρελθόν όμως είχαν τη δυνατότητα να αναπηδήσουν αν θέλετε για να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας να βρει τις συνθήκες που πρέπει να εφαρμόσει όταν ε, ε λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν ούτως ή άλλω απαραίτητη η αλλω απαραιτητη εξυγίανση, αλλά θα πρέπει να βρουν λοιπόν τα κατάλληλα μέτρα που θα τους επιτρέψουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών. Δομικέ αλλαγέ. Αυτό πρέπει να το κάνουν οι κυβερνήσει. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το κάνουμε, ούτε εντολή έχουμε ούτε τη δυνατότητα. Το άλλο ερώτημα που θέσατε. Τις επιπτώσεις του LTRO τραπεζικά συστήματα που αγοράζουν κρατικό χρέος. Ας μην ξεχνάμε ποιο ήταν η κατάσταση πριν. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για απόφαση των τραπεζών και όταν εμείς θέσαμε σε κίνηση τα LTROs, είχαμε ως φιλοδοξία να πάει στην αγορά γρηγορότερα χρήμα. Σήμερα υφιστάμεθα τις επιπτώσεις αυτού του μέτρου, αλλά τα επόμενα χρόνια θα βελτιωθεί η κατάσταση. Οι τράπεζες είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά. Πριν εφαρμοστεί το LTROs, δεν αγόραζαν οι τράπεζες δημόσιο χρέος. Ούτε οι ξένες τράπεζες, ούτε η εθνική τράπεζα κάθε χώρας. Είχαν αποσυρθεί οι ξένοι επενδυτές και οι αγορές οι, οι, των, ομολόγων και όλων των τίτλων ήταν εντελώς κλειστές. Αυτό το οποίο παρατηρείται σήμερα είναι ότι αγοράζουν τα δικά τους ομόλογα, το δικό τους κρατικό κρέος οι τράπεζες και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεπεραστεί. Παρ' όλα αυτά είμαι σίγουρη ότι αυτό το πρόβλημα θα ξεπεραστεί και μόλις ε, οι πιστοτικές αγορές αρχίζουν να λειτουργούν και πάλι θα βελτιωθεί η κατάσταση θα πρέπει να πω ότι από τη θετική πλευρά υπάρχουν δύο θέματα στα οποία θα ήθελα να πιστεί την προσοχή σας. Πρώτα απ' όλα, η κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές τώρα βελτιάνεται βλέπουμε. Στους τρεις πρώτους μήνες είδαμε ότι εκδόθηκαν τίτλοι και χρεόγραφα σε ποσότητα όπως αυτή που είχαμε πέρσι όλο το χρόνο, τους 12 μήνες. Αυτό λοιπόν είναι θετικό. Δεύτερο θέμα θετικό. Αντίθετα με την γενική εντύπωση που υπάρχει τα μέτρα τα οποία προβλέπονται μεταξύ των τραπεζών που έχουν αγοράσει κρατικό χρέος δημιουργούν μία μάλλον θετική κατάσταση. Thank uh, ευχαριστώ πολύ και τώρα για το ECR. Ο Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στην τελευταία μας συνάντηση το Δεκέμβριο σας είπα ότι κάποιοι θέλουν να γίνεται ο Άι Βασίλης της Ευρώπης. Δυστυχώς όμως αυτό ακριβώς κατάληξε να γίνεται. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ρευστότητα τόσο στις τράπεζες σε χαμηλά επιτόκια με αμφιλεγόμενα εγκυμφιλεγόμενες εγγύησεις. Οι τράπεζες χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά για να αγοράσουν εθνικά ομόλογα όμως. Και όχι όμως γίνεται, και μάλλον γίνεται όχι μόνο ο δανειοδότης ε, τελευταίας ε, λύσης, τελευταίας καταφυγής, αλλά ονών. Μόνο χρόνο αγοράσατε, γιατί οι εντάσεις στο ευρωσύστημα μπορεί να επανέλθουν οποιαδήποτε στιγμή. Ιδιαίτερα με εκλεγεί ο κύριος Όλαντ ε, που βρίσκεται σε φάση άρνησης στην Γαλλία. Ερωτώ λοιπόν, μπορεί να με τρίτο LTRO και πότε. Και πότε θα σταματήσετε την πρακτική να αποδέχεστε από εγγυήσεις ε, από τράπεζες, όπως ζήτησε ήδη ο πρόεδρος της Bundesbank, της ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας της Γερμανίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για απάντηση. Νομίζω ότι τα LTRO ήταν αρκετά έγκαιρα και νομίζω ότι ήταν αρκετά επιτυχή τελικά ως ε, ε, δραστηριότητα. Αν τελικά το μόνο που πετύχαμε ήταν να αγοράσουμε χρόνο, που δεν ήταν το μόνο που πετύχαμε, και αυτό όμως από μόνο του θα ήταν τεράστια επιτυχία. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει. 230 δισεκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ στους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Αγορές εντελώς κλειστές. Αυτά τα αποφύγαμε. Αλλά να σας πω γιατί οι τράπεζες δεν δανείζουν. Οι τράπεζες δεν δανείζουν γιατί είτε δεν έχουν χρηματοδότηση ή είτε δεν έχουν κεφάλαιο είτε δεν υπάρχει ζήτηση. Εμείς τι κάναμε. Αφαιρέσαμε τον πρώτο από τους τρεις παράγοντες. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε κεφάλαιο που δεν έχουν οι τράπεζες ενδεχομένω. Και να προσθέσω ευθύ αμέσω ότι έχουμε κάποια τοπικά προβλήματα με τράπεζες. Αλλά γενικά από ό,τι προκύπτει από την αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αυξήσει τα κεφάλαιά τους σε κάποιο βαθμό. Κατά 65% εκτιμάται ότι οι τράπεζες ε, συνάδουν με τους όρους, συμμοφώνονται με τους όρους που τους έχουν οριστεί. Άρα θεωρώ ότι να αγοράζουμε χρόνο δεν είναι κάτι που μπορούμε να το περιφρονούμε δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε έλλειψη κεφαλαίου. Και ιδιαιτέρως, όπω είπα εξ αρχή, δεν μπορούμε εμεί να αντικαταστήσουμε την έλλειψη ζήτηση Για το επόμενο LTRO θα σα δώσω την σταθερή απάντηση που δίνω, ότι ποτέ δεν μπορούμε να δεσμευτούμε εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα για του πράσινου η Πασκάλ. Α, συγγνώμη, κάτι ξέχασα. Κάτι ξέχασα σε ό,τι αφορά την ερώτηση αυτή, που δεν απάντησα. Το θέμα των εγγύσεων. Καταρχάς, γιατί δεν αποδυναμώσαμε, είπατε αποδυναμώσαμε, δεν αποδυναμώσαμε, διευρύναμε την ε, επιλογή εγγύσεων Και γιατί, γιατί θέλαμε να αυξήσουμε τον αριθμό τραπεζών που θα συμμετείχαν στις ε, δράσεις, στα εγχειρήματα αυτά. Καταφέραμε στο τελευταίο LTRO να συμμετάσχουν 800 τράπεζες, 460 εκ των οποίων ήταν γερμανικές. Να έχετε υπόψη ότι η μέση συμμετοχή είναι 70-75. Και γιατί? Γιατί οι εγγυήσεις που ζητούμε θα πρέπει να έχουν κάποια ποιότητα ασφαλώς, αλλά να παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ε, που ουσιαστικά δεν μπορούν να τις παρέχουν οι μικρομεσαίες τράπεζες. Ουσιαστικά λοιπόν είναι οι μεγάλες τράπεζες οι οποίες στρέφονται ε, στα προγράμματά μας, οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες θα διανύμαν τους πόρους αυτούς στις μικρές τράπεζες. Αυτό δεν συμβαίνει όμως τώρα, γιατί η αγορά μεταξύ των τραπεζών έχει κλείσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουν πρόσβαση οι μικρές τράπεζες. Άρα διευρύναμε την επιλογή ε, εγγύησεων. Δεν την αποδυναμώσαμε όμως. Διασφαλίζουμε ότι οι εγγύησεις που συμπεριλαμβάνουμε ανταποκρίνονται στο κίνδυνο που αποδεχόμασταν σε ό,τι αφορά ε, τις προηγούμενες εγγύησεις, στα κουρέματα που αποδεχόμασταν. 53% κατά μέσο όρο περικοπές. Δηλαδή, αν μια τράπεζα ε, φέρνει αυτό το, αυτές τις νέες εγγυήσεις, πρέπει να έχει περίπου το ίμιση του κινδύνου. Αλλά αυτό μπορεί να φτάσει και μέχρι 70%. Άρα θεωρώ ότι ο κίνδυνος, μάλλον η κινδυνολογία σε ό,τι αφορά τις νέες ε, αυτές εγγυήσεις δεν δικαιολογείται. Η Πασκάλα έχει τώρα το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Oui. Καλημέρα κύριε Ντράγκη. Θεωρούμε ότι τα LTRO ήταν απαραίτητα, όπως η μορφή είναι απαραίτητη για έναν άρρωστο, για να πονάει λιγότερο και για να κερδίσει χρόνο. Αλλά δεν ρυθμίζει κανένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα που υπάρχουν και που αναφέρθηκαν από τους διαφορούς συναδέλφους. Θα ήθελα να επανέλθω στο LTRO και στη χρήση αυτών όπως έγινε. Πιστεύω ότι από δημοκρατική άποψη είναι απολύτως νόμιμο να θέλουμε να γνωρίζουμε τι έγιναν αυτά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρηματοδότησαν την πραγματική οικονομία, χρηματοδότησαν τα κρατικά χρέη, κατατέθηκαν στην κεντρική τράπεζα. Αυτή η διαφάνεια του ενός τρεις συγγνώμη, ευρώ πρέπει να αποτελεί συνθήκη για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ορίζει την εμπιστοσύνη που θα έχουμε στην Κεντρική Τράπεζα. Πώς μπορούμε να ζητάμε λιτότητα από τον πολίτη, αν από την άλλη πλευρά θεωρεί ότι ένα τρισεκατομμύριο ευρώ χάθηκαν χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμία διαφάνεια, χωρίς συχνηλασιμότητα. Θέλουμε λοιπόν επίσημους αριθμούς που να μην είναι απλά εκτιμήσεις ορισμένων τραπεζών που ενδεχομένως έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας. Αρνείστε να θέσετε όρους στη χρήση από τις τράπεζες αυτών των ποσών. Γιατί να δώσουμε αυτό το 1 τρισεκατομμύριο, απαραίτητο για τους λόγους που αναφέρατε, αλλά γιατί να μην θέσουμε αντιπαροχές. Κάθε φορά που η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αγοράζει κρατικά χρεόγραφα, ε, έχει δώσει ε, ανταλλάγματα. Αυτό πιστεύω μπορεί να βλάψει την εμπιστοσύνη που έχει το κοινό στην Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Θα σας πω αμέσως ότι πρέπει να συνεχίσετε να εμπιστεύεστε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχουμε στα χέρια μας η εμπιστοσύνη σας στον δικό μας θεσμό. Θα σας παρουσιάσω κάποια επιχειρήματα. Για ποιο λόγο πρέπει να συνεχίσετε να εμπιστεύεστε την ECB. Είχαμε όλες αυτές τις τράπεζες που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση. Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν έχουμε τη γαλλική μετάφραση στο κανάλι 3. Όχι, δεν χάσαμε τη Γαλλία. Είναι ακόμα εδώ. Δεν ξέρω αν μπορούν οι διερμηνείς να πούν κάτι στο κανάλι 3. Νομίζω ότι πρόκειται για μια γενική βλάβη. Τώρα είναι εντάξει. Τώρα ακούγονται. Ναι, ωραία, έχει επανέλθει. Ήταν μια γενική βλάβη. Ζητώ συγγνώμη Μάριο. Ευχαριστώ. Όπως έλεγα, η εμπιστοσύνη σας στο δικό μας θεσμό είναι το μεγαλύτερο πλέον έκτημα που έχουμε στα χέρια μας και θα σας παρουσιάσω κάποια επιχειρήματα ε, υπέρ αυτής της εμπιστοσύνης που πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσετε να έχετε. Τι συμβαίνει με τα LTRO. Τα τριετές LTRO ήταν πρόσδεκτο ως μέτρο που όπως είπα προηγουμένως ανακτά τι, επαναφέρει τη λειτουργία ορισμένων χρηματαγορών για, τους, για τον λόγο ακριβώς ότι ήταν τριετές και όχι τρία-ένα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κατά κάποιο τρόπο διασφαλίζει ότι οι τράπεζες θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τρία χρόνια. Θα έχουν αυτά τα χρήματα για τρία χρόνια. Πρόκειται για μια διασφάλιση ότι δεν θα έχουν έλλειψη ρευστότητα μετά από 6-7 μήνες και πάλι. Αυτό πιστεύω ήταν το σημαντικότερο γεγονός αυτής της δράσης που είναι άνευ για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό που συνέβη είναι ότι εμείς μετά αναρωτηθήκαμε, φαντάζεστε, πού πάνε αυτά τα χρήματα και αυτό που παρατηρήσαμε από το πρώτο ηλτιαρό αμέσως ήταν ότι η ταυτότητα των τραπεζών που δανείζονται ήταν εντελώς διαφορετική από τις τράπεζες που επανακατέθεταν ε, σε αυτό το μηχανισμό. Γιατί συνέβαινε αυτό. Αυτό δείχνει ότι αυτή η ρευστότητα το να, της επανακατάθεσης ε, συμβαίνει σε όλο το σύστημα. Άλλες τράπεζες ε, οι οποίες δεν χρειάζονται αυτή τη ρευστότητα επανακαταθέτουν στο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η πρώτη απόδειξη που είχαμε λοιπόν ήταν ότι αυτά τα ρευστότητα, αυτά τα χρήματα κινούνται μέσα στην οικονομία. Που αυτή ήταν ουσιαστικά η κυρία μας ανησυχία. Αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς πού ακριβώς πηγαίνουν. Ο ισολογισμός της δικής μας Κεντρικής Τράπεζας δεν το δείχνει. Το μόνο που δείχνει είναι ότι εξορισμού, εφόσον δημιουργούμε ρευστότητα, αυτή επανέρχεται στο μηχανισμό καταθέσεων ή σε απαιτούμενα αποθεματικά για να διατηρηθούν τα επίπεδα, αλλά κυρίως ε, στο μηχανισμό καταθέσεων. Χρειάζεται χρόνο για να αυξηθούν τα αποθεματικά, αλλά το πώς και πού καταλήγει στην οικονομία μπορούμε να το μάθουμε μόνο μελετώντας ε, τα ενοποιημένους ισολογισμούς των τραπεζών στις διάφορες χώρες. Αυτό ουσιαστικά παρακολουθούμε. Καθημερινά, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Είναι αδύνατο όμω να παρατηρήσουμε πόσα από αυτά καταλήγουν σε πιστώσει ή σε αγορές κρατικών ομολόγων. Από τα δεδομένα που έχουμε εμεί στη διάθεσή μας πρέπει να συλλέξουμε δεδομένα από τις εμπορικές τράπεζες. Είμαι βέβαιος ότι σε δύο περίπου μήνε ή σε μερικού μήνε θα μπορέσουμε να σα δώσουμε μια πιο ακριβή λεπτομερή εικόνα του τρόπου χρήση αυτών των χρημάτων και πού αυτά καταλήγουν. Έχουμε δει χαρτοφυλάκια ε, τραπεζών για κρατικά ομόλογα να αυξάνονται ειδικότερα για Ιταλικά, Ισπανικά, Ιταλικές, Ισπανικές και άλλες τράπεζες και Γαλλικές τράπεζες. Έχουμε παρατηρήσει αύξηση εκεί. Δεδομένη τη κατάσταση εκείνη τη στιγμή, αυτό ήταν ένα από του λόγου, αλλά τα περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε είναι έμεσα ουσιαστικά. Έχουμε παρατηρήσει εκ νέου άνοιγμα των πιστοτικών αγορών, των αγορών χρηματοδότησης δείτε την έκδοση ομολόγων που έχει λάβει η χώρα μέχρι σήμερα. Όλα αυτά είναι ενδείξεις μιας πραγματικότητας ε, που, για την οποία θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε δύο μήνες ε, κοιτώντας τον ενοποιημένο ισολογισμό. Από άποψη διαφάνειας, οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιοποιηθούν, θα είναι απολύτως καθαρές και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για αυτό το σκοπό. Αλλά ο ισολογισμός μας αυτός καθεαυτός δεν το δείχνει άμεσα. Θέσατε ένα άλλο ζήτημα. Εάν αν διαφωνείτε, πείτε μου το. Θέσατε ένα άλλο ζήτημα. Αναρωτηθήκατε κατά πόσο είναι δυνατόν να ζητούμε από τις τράπεζες ε, να, να μην ζητούμε από τις τράπεζες να πληρούν κάποιους όρους όταν χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα ενώ όταν εμείς ε, χρησιμοποιούμε το S&P ζητούμε από τις χώρες να συμμορφώνονται με αυτούς τους όρους το δεύτερο κομμάτι της δήλωσης αυτής δεν είναι απολύτως σωστό. Εάν είχαμε εμείς πράξει κάτι τέτοιο, μάλλον αφήστε με να πάω λίγο πίσω, θα, έρθω και σε αυτό ναι, που αναφέρετε. Είναι καλές ερωτήσεις αυτές, όντως. Ο λόγος ενεργοποίησης του SMP ήταν ότι οι διάβλοι μετάδοση της νομισματικής πολιτική είχαν φράξει. Είδαμε πέρυσι ότι η νομισματική πολιτική δεν είχε κανένα αποτέλεσμα σε ορισμένες χώρες. Στη συνέχεια θελήσαμε να επαναφέρουμε τις συνθήκες ύπαρξης, τις συνθήκες λειτουργίας αυτών των διαβλών μετάδοσης. Δεν ζητήσαμε απευθείας, είπαμε σε, στις χώρες, σε ορισμένες χώρες, κοιτάξτε, εάν δεν πραγματοποιείστε δημοσιονομική εξυγένση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι απίθανο οι διάβλοι αυτή της νομισματικής πολιτικής να επανενεργοποιηθούν, διότι εμείς μπορούμε να παρέμβουμε αν χρειαστεί, αλλά δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εάν οι αγορές θεωρήσουν ότι εσείς δεν ενεργείτε για να βελτιώσετε την πρόσβασή σα στην αγορά. Για ποιο λόγο δεν ζητάμε παρόμοιους όρους από τις τράπεζες διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί βάσει μια συνθήκη βασισμένη στην ενιαία ελεύθερη αγορά. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατευθύνουμε τις πιστώσεις όπως σε μια προγραμματισμένη οικονομία. Είναι αδύνατο να πράξουμε κάτι τέτοιο. Εξαρτάται, αν μη τι άλλο, οι, οι, οι εθνικές τράπεζες είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Είναι πιο κοντά ε, στις εθνικές τους τράπεζες τιμή, Αν μου επιτρέπετε, δεν υπάρχει ηθικός κίνδυνο με τις τράπεζες ουσιαστικά. Αυτό λέτε. Νομίζω και είμαι βέβαιη ότι τελικά θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, αλλά δυστυχώς ξεπερνάμε τα χρονικά όρια. Ο Γιούγκερ από την Γκουε. <clears throat> Ε, Ευχαριστώ, κύριε Δράγκη. Θα συμφωνήσω με αυτά που σας ρώτησαν ως τώρα, ως πολιτικός, ε, όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους εκλογείς μας, μας λένε πού κατέληξαν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, έχει τεθεί αυτό το ερώτημα επανειλημμένα, αλλά θα ήθελα να σας το τονίσω ότι μας το θέτουν το ερώτημα αυτό οι πολίτες μας. Για πολλούς πολίτες είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι γίνεται. Αυτό στο γερμανικό τύπο παρουσιάζεται ότι αντίστροφα το κοινωνικό κράτος έχει φτάσει στο τέλος τους. Ότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ε, αν αφήσουμε κατά μέρο το κοινωνικό κράτος ε, και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, το δίκτυο ασφαλείας για τους πολίτες, αυτό τι σημαίνει ότι θα σωθούν οι τράπεζες χωρίς να δημιουργηθούν οι όροι ε, και τελικά θα πληρώσει ο πολίτης ε, με αυστηρούς όρους και τελικά θα πληρώσει με τη θέση εργασία του, ε, με την κοινωνική του ασφάλιση, με τη σύνταξή του ο πολίτης. Αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, τουλάχιστον στη χώρα μου, αλλά νομίζω και σε άλλες χώρες. Είναι μια μεγάλη επιβάρυνση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Έτσι γίνεται αντιληπτό τουλάχιστον. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η δική σας θέση, πώς απαντάτε στους πολίτες, θα απαντούσατε στους πολίτες σε αυτά τα βασικά θεμελιώδη ε, ερωτήματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των τραπεζών και του μέλλοντος της δημοκρατίας. Δύο ερωτήσεις κάνατε. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά η ρευστότητα αυτή είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι μαθηματικό, αριθμητικό γεγονός, αλλά στο μεταξύ έχει αλλάξει η ταυτότητα των τραπεζών που εμπλέκονται και έτσι περνάει μέσα από την οικονομία και θα μπορέσουμε να σας πούμε σε τι ε, ποσοστό μετατρέπεται σε πιστώσεις. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το πορτοφόλιο, το χαρτοφυλάκια των τραπεζών σε εθνικέ ε, ομολογίε έχει αυξηθεί. Να σας πω όμως τι τράπεζε ότι αποτελούν ένα απαραίτητο κανάλι για την Ευρώπη. Πάνω από το 80% των πιστώσεων χορηγείται μέσω τραπεζών, σε αντίθεση με τη ΣΥΠΑ, όπου ε, το ποσοστό αυτό είναι 30% και το υπόλοιπο κινείται μέσα από τις κεφαλαίες αγορές. Αν θέλουμε λοιπόν να ξαναξεκινήσει η διαδικασία πιστώσεων, θα πρέπει να περάσουμε από τις τράπεζες. Δεν είμαστε στη ΣΥΠΑ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν το τόνισα επαρκώ, αλλά τα αποτελέσματα της έρευνας για την δανειοδότηση των τραπεζών που θα δημοσιευθούν στις 10 το πρωί είναι ενθαρρυντικά. Δηλαδή, ο κόσμος που παλιά ε, που μάλλον ε, που ζητάει πιστώσεις και δεν τις λαμβάνει, έχει περιοριστεί. Υπάρχουν λοιπόν, ε, υπάρχει κόσμος, μάλλον είναι ακόμα ασθενής, αδύναμη η ζήτηση για πιστώσεις. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι όλο θέμα όμως. Μια δεύτερη ερώτηση απευθύνεται σε μια δήλωση που έκανα για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και ότι είναι νεκρό. Να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Το άρθρο ήταν αρκετά σαφές. Οι αξίες της κοινωνικής συμπερίληψης και της αλληλεγγύης πάντα είναι στην κουλτούρα μου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε βιώσιμο το οποιοδήποτε κοινωνικό μοντέλο. Τα κοινωνικά μοντέλα που βασίζονται σε υψηλό χρέος είναι μη βιώσιμα. Άρα η δήλωση που έρχομαι και κάνω είναι ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ναι, αλλά να είναι βιώσιμο. Γι' αυτό σε κάποιους ε, τομείς της Ευρωζώνης θα πρέπει να διορθωθεί. Αυτή τη δήλωση έκανα. Δεν είμαι κατά της ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το EFD, ο Γκότφριδ. Um, uh, Ευχαριστούμε, κύριε Ντράγκη αν καταλαβαίνω, η δική σας μαχροχρόνια χρηματοδοτική πολιτική είναι να βοηθάτε τις τράπεζες. Σήμερα βλέπουμε ότι δεν μπορούν ούτε η Ιταλική κυβέρνηση ούτε η Ισπανική κυβέρνηση να έρχεται το κεφάλαιο για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις αγορές τους. Από ό,τι κατάλαβα έχουν ε, δοθεί πολλά εκατομμύρια στις, ε, στην ισπανική αγορά. Η 21 δις ε, λείπουν που είναι το μισό από αυτό που χρειάζεται ακόμη να δανειστεί η Ισπανία. Η Ιταλία επίσης χρειάζεται πάρα πολύ, αγορά πάρα πολλών τίτλων και χρεογράφων για να τα καταφέρει. Άρα φαίνεται ότι εσείς δεν θα κάνετε άλλα δάνεια εφέτος. Ίσως ε, μπορείτε να αγοράσετε μέρες και ώρες, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε περισσότερο. Και έχουμε και τους περιορισμούς της συνθήκης του Μάστριτ. Στο άρθρο 1.4 στον κανονισμό σας, δεν ε, είσαστε εσείς κατά της συνθήκης του Μάστρικ, αλλά κατά του άρθρου 104. Εγώ Ήμουνα στην City ε, εδώ και 34, για 34 χρόνια και ποτέ μου δεν είχα εμπιστοσύνη στην ε, και ευρωπαϊκή τα προσωπικά, αλλά την πολιτική της τράπεζας γενικότερα δεν την εμπιστεύομαι. So what's the question? <laughs> Είναι λοιπόν η ερώτηση. Rome Charter. Uh, oh, the answer is yes. Η απάντησή μου είναι ναι. No, no. The answer is yes. Η απάντησή μου είναι ναι. Ούτως ή άλλως. Πρέπει να πω ότι εγώ δεν έχω μπροστά μου του αριθμού που αναφέρατε. Το θέμα όμως είναι το εξή. Θα πρέπει να χρηματοδοτούμε τις τράπεζες ώστε να μπορούν να εξαγοράζουν για ε, οποιοδήποτε ποσό τίτλων και χρεογράφων. Όχι. Οι τράπεζες θα πρέπει να μπορούν ε, για να αποκαταστήσουν ομαλές συνθήκες στην αγορά να είναι σε θέση να αγοράζουν τα δικά τους τα χρέογραφα, αυτά που χρειάζονται. Για να λειτουργεί ομαλά η αγορά. Έτσι πρέπει να ενεργήσουμε. Ευχαριστώ. Ο Χάν Πίτερ από του μία Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Η πρώτη αυτό που προβλέπεται στη Γαλλία, ότι στη Γαλλία ένας από τους δύο υποψηφίους ε, για το προεδρικό αξίωμα είπε ότι θέλει να επαναδραματευτεί το ε, δημοσιονομικό σύμφωνο. Θα προκύψουν ε, αστάθειες στις αγορές. Και πώς προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θεωρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι ήδη υπάρχουν επιπτώσεις. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση για την πατρίδα μου. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις αυστριακές ομολογίες κατά πόσον έχουν αγοραστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε τι ποσοστό και πώς αξιολογείτε την κατάσταση των τραπεζών στην χώρα μου για την μεγάλη έκθεση και σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό από τις ε, εταιρείε αξιολόγηση επιστολεπτικής ικανότητας. Τι, ποιες θα μπορεί να είναι επιπτώσει αυτής. Απάντηση. Αυτό που μας επιφυλάσσει το μέλλον είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα ήθελα να κάνω κάποιες εικασίες Όλοι συμφωνούμε, θεωρώ, ότι οι συμφωνίες αυτές και ο διχασμός αυτός δεν είναι καλός για το ευρώ και ενώ όλοι συμφωνούμε για αυτού, είμαι βέβαιος ότι οι βασικοί παράγοντες της πολιτικής αυτής διαδικασίας όπου οι λαοί είναι κυρίαρχοι, το καταλαβαίνουν και αυτό. Ελπίζω. Είμαι αισιόδοξο και σχετικά βέβαιος ότι πέρα από τις αρχικές διαφορές, πέρα από τις διαφορετικές αρχικές τοποθετήσεις, θα υπάρξει μια συμφωνία από την οποία τελικά θα ενδυναμωθεί το ευρώ και η ευρωζώνη. Αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω αυτό που είπα και στο τέλος της εισαγωγικής μου ομιλίας. Νομίζω ότι πλέον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μακροπρόθεσμα πού οδεύουμε, πού θέλουμε να οδεύσουμε και ποιοι όροι θα πρέπει να πληρούνται, ας αναρωτηθούμε, για να πετύχουμε αυτόν τον απότερο στόχο. Το πιο συγκεκριμένο ερώτημα για το κατά πόσο να αγοράζουμε ή όχι αυστριακούς τίτλους ε, δεν μπορώ να σας το απαντήσω γιατί δεν αποκαλύπτουμε τέτοια στοιχεία. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Περνώντα ξανά στο ΕΛΚ, λενα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την επόμενη Τρίτη θα έχετε κλείσει 1,5 έτος ε, στην θέση σας και θα ήθελα να σας επενέσω γιατί σε αυτό το 1,5 έτος με σαφέ ε, τρόπο καταφέρατε να αποτρέψετε ε, διάφορους κινδύνους και αυτό χρήση επένων. Γιατί ακόμα και τα μέτρα που ελήφθησαν για τις τράπεζες ήταν απαραίτητα επειδή καθυστέρησε τόσο πολύ η πολιτική ανταπόκριση. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σε ό,τι αφορά για τον πληθωρισμό. Είπατε ότι είναι περιορισμένο ο κίνδυνος για τον πληθωρισμό. Αυτό διαφορετικά το εκτιμάει μεγάλο τμήμα της κοινή γνώμης. Πώς το εκτιμάτε ότι είναι χαμηλός αυτός ο κίνδυνος πληθωρισμού. Δεύτερη ερώτηση το γεγονός ότι τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορούν να επιλύσουν τα τροφοδικά προβλήματα των ε, εθνικών τραπεζών. Αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά θα μπορούσατε να παρουσιάσετε τις νέες γραμμές για τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες επί των οποίων αποφασίσατε σε ό,τι αφορά τις ε, εγγυήσεις, τις ασφάλειες που χρειάζεται κάθε τράπεζα. Θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί μια λύση ή τι άλλο χρειάζεται για την τραπεζικό τομέα. Τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο μέλλον θα αποτελεί, ε, θα εξακολουθήσει να αξιοποιεί τη δυνατότητα αγοράς εθνικών ομολογιών στη δευτερογενή αγορά. Και τελευταίο ερώτημα, στην παρούσα φάση στην παρούσα φάση ε, ασχολούμαστε με τις ε, προδιαγραφές στα πλαίσια της Βασιλείας 3. Η περίπτωση της Ελλάδας καταδεικνύει ότι αυτή η μηδενική εγγύηση που χρειάζεται δεν είναι ε, κάτι το οποίο δεν σημαίνει κινδύνους. Θεωρείται ότι υπάρχει κάποια απέτηση που πρέπει να τεθεί σε ό,τι αφορά τα ίδια κεφάλαια. Well, first να σας ευχαριστήσω για αυτό το σπάνιο αγαθό τον έπαινο που μου κάνατε για τις ερωτήσεις, ερωτήσεις σας για τον πληθωρισμό. Αυτό που είπα είναι ότι ο κίνδυνος για τον πληθωρισμό είναι ισορροπημένος. Υπάρχει και ο κίνδυνος αύξησης λόγω των τιμών του πετρελαίου και ε, της ε, έμεσης πρόσβασης, αλλά και ε, κίνδυνο ύφεσης λόγω της αδυναμίας ε, της Ευρωζώνης, με εξαίρεση τη Γερμανίας ενδεχομένω. Ε, οι κίνδυνοι λοιπόν είναι μάλλον ισορροπημένοι σε μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε ο πληθωρισμός ότι πλέον κινείται στο 2,7% και αναμένουμε ότι θα πέσει κάτω από το 2% μέχρι τις αρχές του 2013. υποθέτοντας ε, ότι δεν θα αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων και προϊόντων και με την υπόθεση ότι οι προσδοκίες θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Οποιοδήποτε, ναι, αν θέλετε να κοιτάω κατά πρόσωπο τον ομιλητή στον οποίο απαντάω. Γι' αυτό λοιπόν παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά ενδεχόμενη μεταβίβαση τιμών στους μισθούς και στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς, γιατί θέλουμε να είμαστε βέβαιοι για τη σταθερότητα των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Για το δεύτερο ερώτημα και πάλι. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό το γεγονός ότι κάθε εθνική κεντρική τράπεζα είναι ελεύθερη να αποφασίζει τις εγγυήσεις που θα αποδέχεται. Δεν είναι ορθό αυτό, δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Έχουμε ένα κοινό πλαίσιο Έχουμε κοινού κανόνες και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει από αυτών των κοινών κανόνων και μετά οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες προτείνουν τα μέτρα αυτά. Κάποιος είπε ότι η Ευρωζώνη θα γίνει σαν την ε, αγορά με το ρούβλι της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης. Όχι, δεν ισχύει αυτό, δεν είμαστε κατακριματισμένοι από την άποψη αυτή ο ρόλος των εθνικών κρατικών τραπεζών ήταν πάντα ε, να εκτιμούν τις εθνικές εγγύησεις, αλλά πάντα τηρώντας τους κοινού κανόνες. Για το S&P τώρα. Η αγορά ομολογιών ε, πλέον είναι ένα πρόγραμμα που δεν χρησιμοποιείται για 5-6 εβδομάδες. Αυτό δεν είναι ε, αέναο φυσικά, αλλά δεν θέλουμε να δεσμευόμαστε εκ των προτέρων. Και να σας πω ειλικρινά ότι υπάρχει και ένας άλλος λόγος ε, για τον οποίο δεν κάνουμε δηλώσεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σήμερα, επειδή η αβεβαιότητα για την σημερινή κατάσταση είναι πάρα πολύ υψηλή. Και όπως είπα και την προηγούμενη φορά στην ε, συνέντευξη τύπου, οποιαδήποτε στρατηγική εξόδου είναι πρόορη, Δεδομένη τη σημερινή οικονομική κατάσταση. Επίσης, άλλη μία ερώτηση κάνατε για το μηδενικό ποσοστό κινδύνου για το εθνικό χρέος, για το δημόσιο χρέος. Αυτό δεν είναι η πρόταση του CID4. Δεν το πιστεύουν αυτό πολλά κράτη-μέλη, όπως τα βρείτε από τις τροπολογίες, λέει η Πρόεδρος, αλλά έχει προσελκύσει την προσοχή του Κοινοβουλίου εδώ και κάποιο καιρό σε ό,τι αφορά τον κατακριματισμό. Αν θέλουμε να υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικά επίπεδα κινδύνου για διάφορες χάρες, ασφαλώς θα προκύψει μια πιστοτική αγορά κατακριματισμένη και θα υπάρχει αντίκτυπο σε όλε τι νομισματικέ πολιτικέ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει σοβαρά να το σκεφτούμε. Δεν είμαι βέβαιο ε, κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εντελεχώ μελετήσει το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, θα ήταν ενδιαφέρον να το σκεφτείτε και να μα πείτε. Για το SND ο Λεωνάρντο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγκη, εγώ δεν θα σας κάνω ερώτηση, αλλά κάποιες δηλώσεις και εσείς μπορείτε να μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Η πρώτη δήλωση είναι, διαπίστωση είναι ότι η δημοσιονομική εξυγένση δεν μπορεί να αποφευχθεί. Πολλά εξαρτώνται από τον τρόπο εφαρμογής του και υλοποίησής του. Αυτό σημαίνει να προβλέψουμε μια δυνατότητα προσαρμογή αυτή τη πολιτική εξυγένσης που θα λαμβάνει υπόψη το ρεαλιστικότητα των στόχων ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συνθήκων και των προϋποθέσεων μιας συγκεκριμένης χώρας, ε, ακόμα και χωρών με καλή ρευστότητα. Η δεύτερη δήλωση, η πράξη LTRO είναι επικίνδυνη και ταυτόχρονα ευφυή. Ωστόσο δεν θα είναι επαρκής ε, για να αποφύγει τη μόχλευση των leveraging των τραπεζών όπως αναφέρεται σε μια πρόσφατη έκθεση για την κρίση του διατραπεζικού τομέα. Συνεπώς θα είναι απαραίτητο να βρούμε νέες απαντήσεις και να προωθήσουμε νέες προτάσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Κεντρικών Εθνικών Τραπεζών για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Τρίτη και τελευταία διαπίστωση. Πρέπει να έχουμε ένα μακροπρόθεσμα, όραμα για την Ευρώπη, όπου θα πρέπει να υπάρχει χώρος για νέο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με νέα εντολή, ώστε να μοιράζεται την ευθύνη της οικονομικής διακυβέρνησης. Εάν συμφωνείτε και με τις τρεις αυτές δηλώσεις θα κερδίσουμε χρόνο και εγώ θα δηλώσω απόλυτα ικανοποιημένος. Ευχαριστώ. Πώ ε, ε, Πώς να απαντήσω, στα Ιταλικά ή στα Αγγλικά. Στα Ιταλικά, λέει η Πρόεδρος. λεει ο προεδρος συμφωνω με το 50% των όσων είπατε, <laughs> όπως ε, έλεγε ο γνωστός προπονητής Πρώτον, για τη δημοσιονομική εξυγίανση που υλοποιείται μόνο με φόρους, σίγουρα είναι υπερβολική. Η δημοσιονομική εξυγίανση ιδανικά θα πρέπει να βασίζεται στη μείωση των τρεχουσών δαπανών και μεταξύ αυτών των πιο αντιπαραγωγικών. Όχι λοιπόν να μειώνουμε τις δαπάνες για υποδομές ή επενδύσεις, αλλά τις τρέχουσες δαπάνες. Και όχι να επικεντρωνόμαστε στους φόρους. Συχνά, λόγω του επίγοντος χαρακτήρα ορισμένων περιπτώσεων, αυξάνονται πολλοί οι φόροι. Γιατί, γιατί είναι πιο εύκολο να αυξήσει κανείς τους φόρους παρά να μειώσει τις δαπάνες. Είναι πιο εύκολο από το να μειωθούν οι τρέχοντες λογαριασμοί. Η ύφεση λοιπόν εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η δημοσιονομική εξυγένση όσον αφορά το leveraging των τραπεζών. Να θυμηθούμε, υπάρχουν ορισμένε περιπτώσει τραπεζών σε ορισμένε χώρε τη Ευρωζώνης όπου πρέπει να γίνει leveraging. Διότι έχουν συσσωρεύσει περιουσιακά στοιχεία ενεργητικά λανθασμένα τα οποία βαρύνουν τον προπολογισμό του, τον ισολογισμό του και δυσκολεύουν την δραστηριότητά του. Πρέπει λοιπόν να ρευστοποιηθούν. Το LTRO λοιπόν επέτρεψε να δοθεί χώρος ώστε να γίνει αυτή η ρευστοποίηση assets ενεργητικού με εύλογους όρους χωρίς να προκαλέσει πτώση των τιμών και συνεπώς περαιτέρω απώλειες ε, στα ισοζύγια των τραπεζών. Επέτρεψε δηλαδή να κερδίσουν χρόνο. Το deleveraging ωστόσο είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτές τις δράσεις. Ε, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι δράσεις. Ε, λέμε ότι βοηθάει οι Τράπεζα ζόμπι να επιβιώσουν ενώ δεν πληρούνται οι συνθήκες για να επιβιώσουν. Για το άλλο τώρα, ο Όλε. Σμιτ για το ρόλο της Ευρωπαϊκής και της Κεντρικής Τράπεζας δεν κάνουμε υποθέσεις. Αυτό είναι στα χέρια των νομοθετών. Εγώ πιστεύω, όπως βλέπετε εσείς, έχουμε μία εντολή να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών και ήδη αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Thank you, uh, Mr. Draghi. I have two questions. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Δύο ερωτήσεις και μία έκκληση. Στην προεκλογική εκστρατεία της Γαλλίας όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή και η Τράπεζα και πολλοί οικονομολόγοι λέγουν επίσης ότι αν δεν τα κάνετε όλα λάθος, τουλάχιστον η πλειονότητα των πραξεών σας είναι λαθασμένες. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για την ανάγκη να υπάρχει ανάπτυξη. Πώς σχολιάζετε το ότι δεν κάνετε αρκετά πράγματα για ανάπτυξη. Υπάρχει βούληση να γίνει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο δεν έχει ε, σχέση με αυτό που λέτε εδώ, αλλά αργότερα θα ψηφίσουμε για την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών αλλαγών, αντα, συναλλαγών. Εσείς είστε εδώ ως ε, πρόεδρος ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Σας κάνουμε έκκληση λοιπόν. Εγώ είμαι από χώρα μη ευρωζώνος και κάθε εβδομάδα εμείς και οι πολίτες χώρες προσπαθούμε να καταλάβουμε αν θα είναι επωφελές να γίνουμε μέλος της Ευρωζώνης. Η έκκλησή μου λοιπόν κύριε Ντράγκη σε εσά είναι η εξής. Και φαντάζομαι ότι Είστε ο μόνος Ευρωπαίο στην Ευρώπη σήμερα που προσπαθείτε να εξηγήσετε γιατί είναι εποφελές και πρωταρχική σημασία στην Ευρώπη να έχουμε το ενιαίο νόμισμα. Στη χώρα μου τουλάχιστον πρέπει να πω ότι είναι σχεδόν αδύνατον να προσπαθήσει κανείς να εξηγήσει στη Σουηδία γιατί πρέπει να προσχωρήσει στο ευρώ. Ίσως θα ήταν καλύτερα για την Ευρωζώνη αν η Σουηδία είχε ήδη προσχωρήσει. Ίσως θα ήταν και απόδειξη αλληλεγγύης. Αλλά μην προσπαθείτε να μιλήσετε για τα σημερινά κράτη μόνο και τι θέλετε να κάνετε. Πρέπει να έχετε όραμα και για τις επόμενες δέκα χώρες ευρωπαϊκές που δεν είναι μέλη του ευρώ. Ευχαριστώ. Ακούστε. Λέτε ότι δεν κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ανάπτυξη το δικό μας το καθήκον δεν είναι αυτό. Είναι να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών και μέσω αυτού να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη. Βεβαίως υπάρχουν και δράσεις οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στην οικονομική σταθερότητα. Η νομισματική μας πολιτική επίσης συνεισέφερε και συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Αυτό μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα. Αλλά πώς ξέρετε η ανάπτυξη εξαρτάται και από, πολλούς, από πολλές Πρώτα απ' όλα υπάρχουν θέματα τα οποία είναι θέματα αρμοδιότητες κάθε χώρας και των φορέων που ενεργούν σε κάθε χώρα, των επενδυτών, των πολιτών που πρέπει να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στις αγορές. Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να ανακτήσουν εμπιστοσύνη. Η σταθερότητα των τιμών, η χρηματοπιστωτική πολιτική πρέπει να είναι αντικείμενο εμπιστοσύνης. Αλλά θα πρέπει να ελευθερωθούν και όλες οι ενέργειες που διαθέτει ο καθένας για να ενεργήσουν στην αγορά. Είναι πολύπλοκο το θέμα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι Μόνον όταν επαναδραστηριοποιηθούν όλε αυτέ οι δυνάμει θα βελτιώσουν τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά την ε, φορολόγηση των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν είναι δικό μας θέμα εμείς να εκφράζουμε απόψεις για τους φόρους που προβλέπονται. Αυτό το οποίο είχα πει στο παρελθόν είναι ότι αυτός ο φόρος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι πρακτικής φύσης και να τον υιοθετήσουν όλες οι χώρες. Δεύτερον, διαφορετικά θα έχετε μεταφορά δραστηριοτήτων σε χώρες που δεν εφαρμόζουν αυτό το φόρο. Ή ακόμη χειρότερα, θα περάσετε στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα και εκεί θα γίνονται συναλλαγές που δεν θα βλέπει κανείς τίποτα. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Τώρα, τι λέει η αγορά. Ότι Κάτι τέτοιο θα μειώσει τη ρευστότητα και θα δημιουργήσει ε, καταστάσεις αστάθειας ενδεχομένως και μεγάλων σκαμπανεβασμάτων στην αγορά. Τρίτον, αυτό θα έχει και αυτό είναι δικό μας θέμα, δική μας αρδεότητα, σε κάποια από τα μέσα που χρησιμοποιούμε για τη δημοσιονομική μας πολιτική. Θα πρέπει όλους αυτούς τους περιορισμούς και τα προβλήματα να τα έχετε υπόψη. Και τώρα θα ήθελα να κάνω και μια πιο γενική παρατήρηση. Εμείς προσπαθούμε αυτή την εποχή, δεδομένου ότι περισσότεροι ξένοι επενδυτές και ξένες πηγές χρηματοδότησης έφυγαν από τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, προσπαθούμε να τους προσελκύσουμε για να ξαναγυρίσουν πίσω. Και διαρωτώμεθα αν αυτός ο φόρος είναι ο καλύτερος τρόπος να προσελκύσουμε και πάλι τους ξένους επενδυτές να επιστρέψουν στην Ευρωζώνη. Αλλά αυτές είναι απόψεις κάποιου ο οποίος ούτε είναι εξουσιοδοτημένο να εκφράζει την άποψή του για αυτό το θέμα, ούτε τίποτα άλλο. Η έκκληση τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε γιατί είναι εποφελές να έχουμε ενιαίο νόμισμα. Και ήταν εποφελές τα ωφέλη. Πολλές φορές απαριθμήθηκαν, ατελείωτες φορές στο παρελθόν και εξηγήθηκαν. Σωστά λέτε ότι ίσως δεν είναι κατάλληλη στιγμή να προασπίσουμε την παρούσα κατάσταση, αλλά θα πρέπει να κάνουμε, ε, να δούμε και την προοπτική για το μέλλον. Να δώσουμε αντικειμενικούς ε, μακροπρόθεσμους στόχους στο όραμά μας και να πούμε ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται ώστε να μπορέσει αυτό το όραμα που έχουμε να γίνει πραγματικότητα. Είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν τη στιγμή της υπογραφής ε, της συνθήκης του Μάστερ και όταν Δέκα ή 15 χρόνια πριν κάναμε ένα μεγάλο άλμα προς τα μπρος με το ενιαίο νόμισμα. Και είπανε ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να προχωρήσουμε. Τώρα βρισκόμαστε σε μια παρεμφερή κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα για το ECR Robert Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στην ερώτησή μου θα αναφερθώ σε ένα μικρό ζήτημα για την Ευρώπη, αλλά μεγάλο ζήτημα για ένα κράτος μέλος που δεν είναι η Σουηδία, αλλά δεν είναι πολύ μακριά από τη Σουηδία, τη Λετωνία. Στις αρχές αυτού του μήνα ο Πρωθυπουργό της Λετωνία αναφέρθηκε από την ISP News Agency ότι κατηγορούσε την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παραβιάζει τα κριτήρια του Μάστριχτ περιγράφει τη Λετωνία ως χώρα που λαμβάνει χρηματοοικονομική στήριξη και ότι υπόκειται σε πολιτικές λιτότητας. Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, ουσιαστικά η Λετωνία συγκρίνεται με μία μόνο χώρο που δεν είναι της Ευρωζώνης, είναι ουσιαστικά η Σουηδία. Θεωρώντας λοιπόν ότι ένα ή δύο κράτη-μέλη θα υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην Ευρωζώνη από το 2014. Μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη Λετωνία ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα που είναι έτοιμη να προσχωρήσει στην ε, Ευρωζώνη θα μείνει πιστή στα κριτήρια σύγκλησης ή πρέπει να αναμένουμε κάποια εξαιρετική ή παρά, παράτυπη ή ε, εξαιρετικού είδους προσέγγιση. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω απάντηση ότι θα αξιολογήσουμε τα κριτήρια σύγκλησης όπως κάναμε και στο παρελθόν. Ακριβώς έτσι. Δεν θα υπάρξει επιλεκτική αίτηση ή διακριτική μεταχείριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο ΕΛΚ και στον Μάριο. Μάριο Μόρο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε Δράγκη. Ε, ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων στα ελληνικά κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Τράπεζας. Διότι αντιλαμβάνομαι ότι εσείς μιλάτε τα ελληνικά τόσο καλά όσο μιλάτε και τα γερμανικά. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που σχετίζεται με κάτι που είπατε στην αρχή της ε, παρέμβασής σας που μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ε, όταν αναφερθήκατε στην ευελιξία, σε μια νέα ευελιξία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μου κάνει εντύπωση διότι σε μια εποχή όπου αντιμετωπίζουμε μια τόσο σοβαρή κρίση οικονομική οι κυβερνήσεις ε, είναι πολύ άκαμπτες όσον αφορά τις διερθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, αυτή η ευελιξία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μου φαίνεται το μόνο πραγματικό περιθώριο δράσης το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε την Ήπειρό σε ανάπτυξη. Και μου φαίνεται επίσης ότι η γερμανική κυβέρνηση που είναι ιδιαίτερα άκαμπτη σε θέματα όπως τα ευρωομόλογα ε, φαίνεται να ενδιαφέρεται για αυτή την ευελιξία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χωρίς να θέλω να σχολιάσω αυτή τη δική μου κρίση. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε αυτή την έννοια. Τι είναι αυτή η νέα ευελιξία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν κατάλαβα κάποια πράγματα δεν μου είναι σαφή. Θυμάμαι που μίλησα για ευελιξία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πότε μίλησα. Ε, στην αρχή της παρουσίασής σας κύριε Πρόεδρε mi ε, ε, Μήπως υπήρχε κάποιο θέμα μετάφρασης, διότι εγώ δεν νομίζω ότι χρησιμοποίησα τη λέξη ευελιξία. Μου φαίνεται λίγο παράξενο. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν τη χρησιμοποίησα. Να το ελέγξουμε τώρα. Uh, we'll, we'll, we'll... το ελέγξουμε να δούμε κατά πόσον ε, μπορούμε να το επιλύσουμε και ας περάσουμε στην επόμενη ερώτηση του S&D. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Well, we've got... Let's let's let's go on to to to Liam, <laughs> and and we'll come back on on on the flexibility. Ακούσουμε τον Λίαμ και μετά να επανέλθουμε στην ευελιξία. Alors moi je suis élu de France. Ευχαριστώ, Σάρων. Εγώ είμαι Γάλλος, ε, αλλά δεν θα αρχίσω να κατηγορώ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν ασχολείται με την ανάπτυξη δεδομένων των μη συμβατικών μέτρων που πήρατε, όπως υπογράμμισε ο φίλος μου ο Κομφάου το πραγματικό ζήτημα είναι η στρατηγική τόνωση τη ανάπτυξη σήμερα στην Ευρώπη. Όπω είπατε και εσεί, ο ίδιο δεν εξαρτάται μόνο από την νομισματική πολιτική, αλλά και από το σωστό μείγμα πολιτική. Αυτό θα είναι το αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευση τη συνθήκη ε, που θα ζητήσει η Γαλλία σε περίπτωση αλλαγή κυβέρνηση τη 6 Μαου. Η γραμμή που φαίνεται να υπερασπίζεστε ε, θα την ονόμαζα γραμμή Ευρωπαϊκού Ταμείου όπως εξηγήθηκε, γνωρίζετε το οικονομικά έγγραφα, αναφέρομαι στα περίπτωση Μακμίλαν. Αυτή η γραμμή λοιπόν συνίσταται στην υποστήριξη μιας νομισματικής πολιτικής επεκτατικής τελικά και περιοριστική απόψη δημοσιονομική μαζί με πολιτικές διαρθρωτικής μεταρρύθμισης υλοποιείται εδώ και ένα χρόνο με ελάχιστα καλά αποτελέσματα διότι μας ανακοινώνεται για του χρόνου μια ύφεση στην Ευρωζώνη. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι επενδύσεις ε, δεν ε, βοηθούν, δεν ε, καθοδηγούνται από τις πολιτικές, αλλά καθοδηγούνται από τη ζήτηση. Οι, ουσιαστικά οι επιχείρησεις δεν ζητούν πιστώσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η νομισματική πολιτική σε μια περιοχή ύφαση. Μπορούμε σήμερα να μην έχουμε δημοσιονομική πολιτική. Μου λέτε ότι δεν έχουμε περιθώριο χειρισμού. Αλλά το γνωρίζετε και αναφερθήκατε προηγουμένως ότι υπάρχει μια διάκριση που λέει ο Κέινς στην Επιτροπή Μακμίλαν μεταξύ του προπολογισμού λειτουργίας που πρέπει να είναι ισορροπημένος και του προπολογισμού κεφαλαίου που μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο δανεισμού για να χρηματοδοτήσει στο μέλλον ε, τις επενδύσεις με τρόπο αντικυκλικό. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ποια θα είναι η δική σας στάση σε περίπτωση που αλλάξει η κυβέρνηση η Γαλλία και προτείνει να εξαιρέσουμε από τον υπολογισμό των δημοσίων ε, ελλημάτων τις, επενδυτικές, τις δημόσιες επενδυτικές δαπάνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως είπα, είμαι σίγουρος ότι οι παράγοντες της πολιτικής αλλαγής θα βρουν μια κοινή γραμμή για να υπερασπίσουν το ευρώ. Ας μην ξεχνάμε ειδικά για να απαντήσω την ερώτησή σας ότι το ζήτημα του εξαίρεση των κεφαλαικών δαπανών από τη λογιστική του Μάστριχτ συζητήθηκε την εποχή της συνθήκης του Μάστρεχτ το 1992 ξανασυζητήθηκε την εποχή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και στις δύο περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι ήταν τρομακτικά δύσκολη έννοια, τρομακτικά διφορούμενη έννοια, δύσκολο να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα μια τέτοια εξαίρεση. Απλά σα δίνω ένα ιστορικό στοιχείο, μια ιστορική υπενθύμηση επί του θέματος. Έτσι έχει ιστορικά το ζήτημα. Ας δούμε τώρα τι θα κάνουν ή όσοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ε, ενώ ωστόσο πράγμα θα ήθελα να προσθέσω λέτε ότι εδώ και ένα έτος έχουμε συρρυκνωτική δημοσιονομική πολιτική. Αυτό δεν ισχύει για ορισμένες χώρες. Κάποιε χώρε σημειώνουν μεγάλη πρόοδο αυτή τη στιγμή. Αυτή η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική ξεκίνησε να υλοποιείται πολύ πιο πρόσφατα από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του περσινού έτους. Σε άλλες χώρες έχετε απόλυτο δίκιο. σε άλλες χώρες είναι και πάνω από ένα έτος. Συνεπώς είναι ετερογενής η κατάσταση. Μπορώ να το πω αυτό. Δεν είναι απάντηση στην ερώτηση βέβαια. Ναι βεβαίως, λέει ο Πρόεδρος. Θα σας δώσω τα αποτελέσματα της έρευνας δανεισμού των τραπεζών του 2012 που μόλις δημοσιεύτηκε. Συνολικά τα αποτελέσματα είναι θετικά. Η μεγάλη επιτάχυνση των περιορισμών το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο πέρυσι αναστράφηκε. Αναμένεται περισσότερη χαλάρωση των τραπεζών στο δεύτερο τρίμηνο. Σημείωσαν οι τράπεζες βελτίωση όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, σε όλες τις κατηγορίες χρηματοδότησης, ειδικότερα για τα κρατικά ομόλογα και τις χρηματαγορές παρομοίες στις προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2012 αναμένονται ε, κάποιες βελτιώσεις. η έρευνα καταδείκνει ότι κατά την αντίληψη των τραπεζών οι επιπτώσεις και αυτό μας απαντάει μια από την ερώτηση της ε, κρίσης κρατικού χρέους ε, στις ε, συνθήκες χρηματοδότησης έχει μειωθεί. Θα σας, θα σας προειδοποιήσω ωστόσο χρειάζεται κάποιος χρόνος για να το αντιληφθούν αυτό οι επιχειρήσεις δεδομένης της χαμηλής ζήτησης για πιστώσεις. Θεώρησα ότι πρέπει να σας αναφέρω αυτές τις ειδήσει. Αυτή την είδηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ψάχνουμε ακόμα να βρούμε πού είπατε τη λέξη ευελιξία. Δεν το βρήκαμε ακόμα. Η επόμενη ερώτηση τώρα από το ΕΛΚ από την Κορίν Βορτμαν Κόλ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Ντράγκη. Θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω ότι θαυμάζω τον ε, τρόπο με τον οποίο διευθύνεται την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε καιρούς κρίσης και θα συνεχίσω στα Ολλανδικά επειδή είμαι από την Ολλανδία θα ήθελα να σας ε, επιστήσω την προσοχή σε αυτά που είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα κράτη-μέλη, μάλλον δεν μπορεί να αντικαταστήσει την λειτουργία των κρατών μελών που δεν ε, δίνουν αποτελέσματα. Το Σεπτέμβριο ασκήθηκε έντονη κριτική. Τότε ε, δεσμεύτηκαν σε αυστηρούς όρους στα πλαίσια του Six-Pack και του 2-Pack σε ό,τι αφορά αυστηρούς όρους για την ανάπτυξη και το δημόσιο χρέος. Αλλά τώρα φαίνεται ότι η Γαλλία και η Ολλανδία δεν είναι διατεθειμένες να κάνουν αυτά που πρέπει και η πολιτική κατάσταση τα επιδεινώνει όλα αυτά. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να τα εξετάσουμε αυτά λίγο πιο ενδελεχώς. Τι αναμένετε ότι θα συμβεί στη Γαλλία και στην Ολλανδία σε τέτοιους καιρούς κρίσης και τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πώς μπορείτε να ασκήσετε νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια αν τα κράτη-μέλη πολύ απλά δεν ε, διατίθενται να τηρήσουν τα όρια, τους όρους σύγκλησης. Τι σημαίνει αυτό για σας και σε περίπτωση που θα ενταθούν ε, οι τριβές. Είσαστε πολύ διστακτικός για να παρέμβετε, δηλαδή θα πρέπει να προκύψει ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης ε, με την υποστήριξη του φορολογούμενου της Ολλανδίας Κάνατε εικασίες πριν από λίγο για το τι πριν από λίγο και είμαι πολύ περίεργη να μου πείτε τι σημαίνει αυτό για την κατάσταση στη Γαλλία και στην Ολλανδία. As, uh, as I said, uh, as I... Όπως είπα και προηγουμένως, σας ευχαριστώ καταρχάς για τους επένους. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι εύκολο το ζήτημα αυτό, γιατί καταρχάς ε, θα εξαρτηθεί από πολιτικά αποτελέσματα που δεν έχουν ακόμα ε, διαμορφωθεί, από πολιτικές αποφάσεις που δεν έχουν ε, ακόμα ληφθεί. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να προκαταβάλω και τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις και να βγάλω κάποιο πόρισμα. Αυτό που μπορώ να πω ωστόσο γενικά είναι ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αξιόπιστο χώρο σε ό,τι αφορά την σταθερότητα των τιμών, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την ε, ανάπτυξη. Αυτό όλοι οι παράγοντες θα πρέπει να το έχουν κατά νου. Ε, μια, ένας αξιόπιστος χώρος ε, σταθερότητας τιμών, δημοσιονομική σταθερότητας και ανάπτυξης. Αν δεν συντρέχουν αυτοί οι όροι, όλοι αυτοί θα μειωθεί η αξιοπιστία της Ευρωζώνης και βασιζόμαστε, όπως όλοι οι χώροι κοινού νομίσματος, ε, βασιζόμαστε το κατά πόσο είμαστε αξιόπιστοι στον υπόλοιπο κόσμο. Έως τώρα, εν γέννη, με κάποιες πρόσφατες ε, εξαιρέσεις, αυτοί οι όροι ε, έστεκαν, υπήρχαν. Υπήρχαν φυσικά παρεκκλήσει, υπήρχαν κάποιες εξαιρεσει, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αξιοπιστία μας σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Για την ε, αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πω το εξής. Συνίσταται στην ικανότητα να αντιδράσει στα προβλήματα που υπάρχουν. Τίποτε δεν εμποδίζει στη συνθήκη την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να ακολουθήσει την κατάλληλη διαδικασία. Εκεί λοιπόν, σε αυτό έγκυται η ε, αξιοπιστία. Τώρα, όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως έχει σχέση με την ε, λειτουργία του Ευρωζώνης διότι έχει σχέση με τις νομισματικές πολιτικές που πολλές φορές ήταν πάρα πολύ χαλαρές εκ μέρου των κρατών μελών και έτσι δεν μπόρεσε να υπάρχει, ε, να δημιουργηθεί η απαραίτητη ανταγωνιστικότητα. Έχει λοιπόν και μια ευρωπαϊκή διάσταση στο ιδιωτικό χρέο. Δεν πιστεύετε ότι ε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το fiscal compact, δηλαδή το δημοσιονομικό σύμφωνο, δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένα financial compact, ένα ε, χρηματοπιστωτικό σύμφωνο για να μπορέσουν να επιληθούν διάφορα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεδομένου ότι, επαναλαμβάνω, το, ιδιωτικό χρέος έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο όλο το σύστημα λειτουργεί στην Ευρώπη. Δεύτερον, ένα σχόλιο. Μιλήσατε για τον περίφημο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και την προσέλκυση επενδυτών. Πρόκειται όμως για το εξή. Γιατί οι καταναλωτές Τες χρηματοπιστωτικών προϊόντων και η χρηματοπιστωτική αγορά θα πρέπει να έχουν πλεονεκτήματα συμπληρωματικά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Διότι πιστεύω ότι οι, όλοι οι καταναλωτές και όλες οι παραγωγικές βιομηχανίες, όλοι το τομείς της οικονομίας θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση στην Ευρώπη για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη. Σωστά είπατε ότι έχουμε το Fiscal Compact, αυτό το σύμφωνο, και αυτό το οποίο σκέφτομαι τώρα είναι να έχουμε μια, ένα growth compact, ένα σύμφωνο ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο προβλεπόταν στο six pack. Θα πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν και να το six pack αυτό, αυτά τα έξι μέτρα φερρυπή να τα κάνουμε σύμφωνο. Αυτό που χρειαζόμαστε και το είπα προηγουμένως στην αγωγική μου παρατήρηση είναι να προχωρήσουμε με την ε, ε, δημοσιονομική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έλεγα ότι είναι μία περαιτέρω θα έλεγα ότι μία περαιτέρω πηγή του κατακαιρματισμού σήμερα είναι η διαφορετική τρόπη με την οποία οι εθνικές εποπτικές αρχές εφαρμόζουν τους κοινούς κανόνες. Τώρα, ε, είπατε για δημοσιονομικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει το τραπεζικό σύστημα. Συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει εδώ να υπάρχουν πλεονεκτήματα επιμέρους για κάποιον τομέα της οικονομίας. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ίση μεταχείριση την οποία μέσω φορολογικών μέτρων θα πρέπει να επιτύχουμε για όλους. Κανένας δεν θα πρέπει να υποφελείται περισσότερο με συστήματα ειδικά φοροπαλλαγών. Δεν θα πρέπει κανένας να ευνοείται περισσότερο από τους άλλους. Και αναφέρουμε στον τραπεζικό τομέα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλώς ορίσατε κύριε Ντράγκη. Μιλήσατε σήμερα το πρωί για το μέλλον και για το σύμφωνο ανάπτυξης δεν θέλω να μου απαντήσετε απαραίτητα, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε τη γλώσσα της λιτότητες. Εγώ διευθύνα τέσσερα ε, δημοψηφίσματα υπέρ της Ευρώπης στην Ιρλανδία και αυτό αποτέλεσε τεράστιο παθητικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το δημοσιονομικό νομισματικό ταμείο. Δεν έχουμε καμία... Ε, αντίληψη του τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες. Πρέπει να εξηγήσουμε τη λιτότητα, πρέπει να εξηγήσουμε τους σκοπούς. Πρέπει να ακούσουμε περισσότερα για θέσεις εργασίας, για ελπίδα, για το μέλλον. Έχουμε βαρεθεί την λιτότητα, σας παρακαλώ, όσον αφορά τη γλώσσα. Θεωρώ ότι πρέπει να δείχνει περισσότερη κατανόηση για το λαό. Στην Ιρλανδία έχουμε το δύο λέξεις, trust και confidence για την εμπιστοσύνη. επανέρχεται σιγά σιγά η εμπιστοσύνη με την αύξηση των επενδύσεων στην Ιρλανδία, αλλά οι ταμιακές ροές μειώνονται. Έχουμε τεράστιο ιδιωτικό χρέος το οποίο συμπεριλάβαμε στο δημόσιο ισοζύγιο. Και θέλω να σας ρωτήσω όσον αφορά τις ταμιακές ροές. αναμένεται ότι υπό όλε αυτέ τι συνθήκε ότι μπορούμε να εξακολουθήσουμε να πληρούμε τι συνθήκε του Promissory Note. Μήπω πρέπει να το επαναδιατυπώσουμε, να έχουμε κάποια ευκαιρία για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ώστε αυτέ οι ταμιακέ ροέ να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και να επανέλθουμε σε ανάπτυξη. Αυτό που είδαμε στην Ιρλανδία είναι μια ισχυρή δέσμευση για την υλοποίηση των προγραμμάτων των πολιτικών. Η στάση της ελλανδικής κυβέρνησης σήμερα εστιάζεται ε, για την έβρεση μιας βιώσιμης ε, οδού και για να συνεχιστούν ε, οι μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Παρ' όλα αυτά παραμένουν προκλήσεις. Η επαναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα στην Ιρλανδία χρειάζεται να ολοκληρωθεί τα ισοζύγια των τραπεζών πρέπει να ενισχυθούν και πρέπει να ενισχυθεί και η πρόσβαση της Ιρλανδίας στις αγορές. Πιο συγκεκριμένα για τη δική σας ερώτηση του κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα σκοπεύει να κάνει οτιδήποτε σε σχέση με τους σημερινούς όρους ε, συμβάσεων. Υπάρχουν αυτοί οι όροι και είναι αυτοί που είναι. Έχουμε κάνει μερικά βήματα. Θα συνεχίσουμε να προβληματιζόμαστε επί του ζητήματος στο άμεσο μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε αυτούς τους όρους. Ευχαριστώ. Thank you now for the Σας ευχαριστούμε, ο Πίτερς είπε για την ε, Σολστές. Κύριε Πρόεδρε, Ράγκη. οι απαιτήσει της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Σύστημα εκτιμούνται στο διπλό των δαπανών του γερμανικού προϋπολογισμού που εξοργίζει πάρα πολλούς. και θεωρείται ότι αυτό αποτελεί απόρρια ενός κρατούς μέλους. Τους τελευταίους μήνες αυξάνεται όμως ο κίνδυνος στην Ευρωζώνη και ένας Ευρωπαίος καθηγητής ποινικού δικαίου, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε για ανελικρίνεια. ότι υπάρχει ανισορροπία σε ό,τι αφορά ε, το σύστημα πληρωμών. Πρόκειται για λεπτομέρειες ή πρόκειται αυτό να προκαλέσει περαιτέρω προκλήσεις στην Ευρωζώνη. Thank you. Uh, no, I think the target Νομίζω ότι οι ισολογισμοί του στόχου 2 αποτελούν ένα εξαιρετικό σύστημα του συστήματος πληρωμών. Αποτυπώνουν ουσιαστικά διατραπεζικές και διεθνικές ροές υπό φυσιολογικούς όρους δεν θα βλέπαμε τόσο υψηλές ε, πληρωμές υπέρ μίας χώρας και ουσιαστικά να είναι τόσες πολλές άλλες χώρες, ή πιο πολλές άλλες χώρες αφού τη μία χώρα. Άρα ε, ο στόχος 2 ε, και αυτές οι ανισορροπίες αποτυπώνουν και είναι σύμπτωμα μιας ε, υποκείμενης κατάστασης. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα, γιατί αποτελούν τμήμα μόνο του συστήματος πληρωμών. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υποκείμενη ασθένεια. Και η υποκείμενη ασθένεια σχετίζεται με το διαφορετικό επίπεδο ανταγωνιστικότητα στις διάφορες χώρες διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, πρόσβαση στην αγορά μεταξύ των διαφορετικών χωρών. Και ως εκ τούτου δημοσιονομική σταθερότητα, βιωσιμότητα και ανάπτυξης στις ε, διαφορετικέ χώρες. Να μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από πέντε χρόνια οι ισορροπίε αυτές δεν προκαλούσαν οποιαδήποτε ανησυχία. Θα δούμε λοιπόν ότι αν γίνει ε, δημοσιονομική εξυγίανση στις ε, χώρες που χρωστάνε. Αν ανακάμψει η ανάπτυξη, αν ανακάμψει η αξιοπιστία, θα δούμε λοιπόν ότι αυτές οι ενισορροπίες στον ε, τομέα, στον στόχο 2, θα επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και να σας πω ειλικρινά, το να θεωρήσει κανείς ότι είναι επικίνδυνες για τους πιστωτές δεν στέκει, γιατί είμαστε μια ένωση και είμαστε όλοι μαζί. Σε ένα σύστημα πληρωμών τα διάφορα μέρη δεν έχουν ε, μεγαλύτερο κίνδυνο, δεν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αν παραμείνουν μαζί από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάρκος από το ΕΛΚ. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε Δάγκη. Στα εισαγωγικά σας σχόλια μιλήσατε για μια οικονομική πολιτική συνεργασία στο ιστορικό της Ευρωζώνης. Αλλά τα πράγματα έχουν ως εξή. Και στο ιστορικό κάποιων κρατών μελών έχουμε μεγάλα, μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ε, διαφορές παρά το γεγονός ότι στα κράτη-μέλη ασκείται μία ενιαία οικονομική πολιτική και στο Βέλγιο, για παράδειγμα, μεταξύ Βορρά και Νότου, στην Ιταλία μεταξύ Βορρά και Νότου, στην Ισπανία και μπορώ να συνεχίσω. Στην Ουγγαρία μεταξύ Ανατολή και δύση υπάρχουν διαφορές. Ας κοιτάξουμε όμως σε επίπεδο ευρωζώνης οι σταθεροποιητέ που οδηγούν σε κατάργηση των διαφορών ακριβώς αυτών. χρειάζονται και μια ενίσχυση ε, ευρωπαϊκή διαμόρφωση των ε, παραγόντων αυτών σταθεροποίησης. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, ποια είναι η γνώμη σας από αυτού. Thank ε, Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να με κατανοήσετε σε αυτά που λέω ως εξής. Και το έχω πει πολλές φορές αυτός. Είμαστε σε μια ένωση, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε συγχρόνως. Πρέπει να έχουμε δρόμο που θα ακολουθήσουμε και σημείο άφηξης. Και θα πρέπει να δούμε πριν να αρχίσουμε αυτό το δρόμο, πριν να προχωρήσουμε, τι είδους μέτρα πρέπει να λάβουμε. Και ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι κάθε χώρα μπορεί από μόνη της να κατορθώσει κάτι. Αυτό ήθελα να πω όταν είπα ότι πρέπει να εξηγήσουμε καλά ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή πριν να προχωρήσουμε. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να μην μείνουμε στάσιμοι και στατικοί στο σύστημα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να οπλιστούμε με ό,τι μέτρα μπορούμε για να προχωρήσουμε. Είμαι πεπισμένος και η πραγματικότητα των τελευταίων μηνών μου δίνει την πεποίθηση ότι είμαι σωστός. Θα πρέπει να είμαστε διαρκώς εν κινήσει. Ευχαριστώ. Ο Γκούναρ Χόκμερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκτός από το γεγονός ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Βίλι Σμίθ τον ε, συμπολίτη μου, για τον ε, φόρο αυτό των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, γιατί είναι παράξενος τρόπος τον οποίο ε, θέλουμε να ενεργήσουμε σημερινές αγορές, θα πω το εξής. Κάτι που είδαμε στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι ότι δεν δημιουργείται ε, κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη βλέποντας πώς έχουν τα ελλείμματα τα σημερινά. Όντως, ε, εάν το δημόσιο έλλειμμα ήταν η λύση του προβλήματος, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Και θα ήθελα να το συζητήσω αυτό μαζί σας, διότι στα πλαίσια του bailout, των PCIs που προβλέπονται, βοηθούνται οι οικονομίες. Και όπως είπατε, είναι σημαντικό όχι μόνο να αγοράσουμε το χρόνο, αλλά και πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε. Αγοράζοντας χρόνο, σημαίνει ότι καταβάλλεται ένα κόστος. Το θέμα λοιπόν είναι, ε, με αυτό που κάνουμε θα βελτιωθεί η κατάσταση ή μήπως ε, τα πράγματα είναι χειρότερα. Πιστεύετε ότι ο χρόνος που αγοράζουμε αγοράζεται για να βελτιώσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητά μας να χειριστούμε τις ανισορροπίες που υπάρχουν στις διάφορες οικονομίες. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό που κάνουμε ε, είναι σωστό. Νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα είπατε. Το ερώτημα είναι το εξής. Οι χώρες και οι τράπεζες σήμερα είναι σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το διαρθρωτικό που έχουν, το τραπεζικό που έχουν, το αναπτυξιακό που έχουν. Και αν δεν είχαμε LTROs θα ήταν καλύτερα οι τράπεζες, αλλά θα είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης. Όταν αποφασίσαμε λοιπόν να ενεργήσουμε τον τρόπο, ενεργήσαμε ήταν όχι για να, εάν θέλαμε να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες και να έχουμε πρόβλημα στα δημόσια οικονομικά όλων των χωρών, δεν θα είχαμε επιτύχει την καλύτερη λύση για τα προβλήματά μας, ούτε για τις χώρες, ούτε για τις τράπεζες. Πιστεύω λοιπόν ότι έτσι πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα. Και σήμερα το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο των κυβερνήσεων και των τραπεζών που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν και να αποδείξουν ότι θα το κάνουν. Όπως σας είπα, οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες, κάποιες από αυτές τουλάχιστον, ε, μας αποδεικνύουν ότι όντως χρησιμοποιούν το χρόνο που αγόρασαν με κάπως παραγωγικό τρόπο ο καθένας ανάλογα με τα αυτά που μπορεί να κάνει. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιου είδους αποδείξεις και μαρτυρίες. Αν όμως έπρεπε εγώ να κρίνω τα LTROs, έτσι θα τα έκρινα. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση του Ζαν Πολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα προβλέψει να πάρω το λόγο, αλλά παραμένει μια χρονοθυρίδα διαθέσιμη Έλεγα λοιπόν ότι δεν είχα προβλέψει να μιλήσω, αλλά υπάρχει χώρο, συνεπώ θα το πράξω. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας πω ότι εκτίμησα ιδιαίτερα το σθένος και το θάρρος των όσων λέτε. Θέλω να σας θέσω μια ερώτηση κάπως ε, προκλητική και σχετική με όλα αυτά. Στις σημερινές συζητήσεις ε, μιλάμε για αύξηση, για λιτότητα, για ανταγωνιστικότητα, όλο και περισσότερα. Εν τέλει αυτό που αναρωτιούνται οι συμπολίτες μας είναι πώς θα γίνει η αύξηση, πώς θα επιτευχθεί καλύτερη ανταγωνιστικότητα, πώς θα επιτευχθεί λιγότερη λιτότητα και δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη απάντηση για αυτές τις ερωτήσεις. Κάθε φορά συζητάμε τα ίδια. Όλο τα ίδια, αλλά ο πολίτης δεν το αντιλαμβάνεται κοιτώντα τα πρόσφατα αποτελέσματα των ερευνών. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι μπορούμε να πούμε πιο συγκεκριμένα πέραν από τα απλά λόγια της αύξησης, της ε, μικρότερης λιτότητας και της καλύτερης ανταγωνιστικότητας. Ευχαριστώ. Well, I I answer, but... Uh, Μακάρι να ήξερα την απάντηση. Συλλογικά πιστεύω βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Βρισκόμαστε, πιθανώς διερχόμαστε στην πιο δύσκολη φάση της διαδικασίας, όπου η λιτότητα, ουσιαστικά η δημοσιονομική εξυγίανση, έχετε δίκιο, η δημοσιονομική εξυγίανση λαμβάνει αυτή τη στιγμή χώρα και τώρα αρχίζει κατά κάποιο τρόπο να φέρνει αποτελέσματα μετά τους περιορισμούς. Δεν έχουμε δει ακόμα αυτά τα ωφέλη αλλά ταυτόχρονα είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να επιμείνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κάθε χώρα είναι διαφορετικές. Δεν μπορούμε να γράψουμε ένα πρότυπο το οποίο θα ίσχυε για όλες τις χώρες. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πλήττουν συγκεκριμένα κατεστημένα συμφέροντα. Διαφορετικά θα είχαν εφαρμοστεί πριν από πολύ καιρό. Αυτά τα κατεστημένα λοιπόν συμφέροντα που πλήττονται οδηγούν ε, ε, τις κοινωνίες σε τεράστιες αλλαγές και από μόνο του αυτό αποτελεί πηγή πόνου. Βρισκόμαστε λοιπόν στα μέσα του ποταμού που διαβαίνουμε και η μόνη απάντηση σε αυτό είναι ότι πρέπει να εμείνουμε και ότι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκό για αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο λεπτά. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Και ο κύριος Γκολτιέρη ζήτησε το λόγο, να του δώσω το λόγο για μια σύντομη ερώτηση. Ευχαριστώ. Μεταλλεύομαι και εγώ το διαθέσιμο χρόνο. Ήθελα να επανέλθω σε κάτι πολύ σωστό που είπατε σε σχέση με τα ζητήματα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Το πρόβλημα είναι η ζήτηση, είπατε. Μα αν το πρόβλημα είναι η ζήτηση, πώς υπό τις παρούσες συνθήκες, ε, πώς θα μπορούσαν οι ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, να μας εμποδίσουν να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο ύφεση που θα μπορούσε να επιδεινωθεί. Μήπως θεωρείτε καθαρά από άψη αναλυτική ε, ε, καθορίσατε ήδη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά κάνοντας μια ανάλυση μήπως είναι ανεπαρκής ε, η απάντηση με μια αποτελεσματική νομισματική πολιτική και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, δεδομένου του ενδεχόμενου ύφαση. Έτσι λοιπόν τίθε το ζήτημα της ε, ζήτησης και των ε, επενδύσεων και είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο δεν μπορούμε πια να αποφύγουμε. Ναι, η ανάπτυξη, απάντηση, η ανάπτυξη δεν οφείλεται μόνο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και στη γενικότερη ζήτηση στην καθολική ζήτηση η οποία έχει παραμείνει αρκετά σταθερή ουσιαστικά οι εξαγωγές μας αυξάνονται και οι εξαγωγές ε, της περιοχής της Ευρωζώνης. Οφείλεται επίσης το γεγονό ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά. Είναι αρνητικοί οι δείκτες εδώ και πολύ καιρό. Εάν κάποιο ε, ήθελε να δημιουργήσει συζήτηση αυξάνοντα τα ελλείμματα, ε, έχουμε τόσο ψηλά ελλείμματα που αναρωτιέται κανεί γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Πράγματι, υπάρχουν χώρε, έχετε υπόψη σα, με υψηλό έλλειμμα και χαμηλό. Με υψηλά και χαμηλά επιτόκια. Και ποτέ δεν σημείωσαν ανάπτυξη. Το ποσοστό ανάπτυξή του, ο συντελεστή ανάπτυξή του είναι flat, είναι σταθερό όποιε και αν ήταν οι δημοσιονομικέ συνθήκε. Η ρίζα λοιπόν αυτή τη έλλειψη ανάπτυξη βρίσκεται αλλού. Και αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουμε πριν μπορέσουμε να πούμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε χώρο στη νομισματική και ε, δημοσιονομική πολιτική, διότι χώρες που απόλυσαν ανταγωνιστικότητα τα τελευταία χρόνια έτσι έκαναν. Δεν είναι ότι την έχασαν για ένα χρόνο, οπότε μπορεί κάποιο να προσδιορίσει μια συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική ω πηγή τη έλλειψη Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία διήρκησε 10 με 15 χρόνια για ορισμένε από αυτέ τι χώρε όπου ε, υλοποιήθηκαν παντός είδους πολιτικές, επεκτατικές ή όχι, ε, ανάπτυξη ή όχι. Και παρόλα αυτά δεν σημειώθηκε ανάπτυξη. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην παρουσία στιγμή. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Ορισμένες οδηγούν σε βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη αλλά άλλες μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη, διότι αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων μηχανισμών της κοινωνίας και διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η ζήτηση όμω οφείλεται επίσης και στην παγκόσμια ζήτηση και από το επίπεδο των επιτοκίων. Το άλλο που μπορεί να αλλάξει είναι ότι αναμφίβολα ένα μεγάλο μέρο τη τρέχουσα κρίση οφείλεται στο γεγονό ότι το κόστος του κινδύνου αυξήθηκε υπερβολικά μετά την κρίση. Συνεπώς, σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχει βούληση επένδυσης, υπάρχει βούληση επένδυσης αλλού. Θα πρέπει να δράσουμε έτσι, ώστε αυτό το κόστος του κινδύνου να επανέλθει όχι στα παλιότερα επίπεδα, διότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, αλλά σε επίπεδα τέτοια ώστε να μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις και ένα κλίμα βεβαιότητας, ένα περιβάλλον βεβαιότητας, αξιοπιστίας, βεβαιότητας και αξιοπιστίας όσον αφορά τους θεσμούς και τότε θα δούμε το κόστος του κινδύνου θα μειωθεί. Thank you very much ε, indeed. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα είναι ενημερωτικό και ενδιαφέρον να σας έχουμε πάντα. Και παρά τις ε, επικρίσεις που ακούστηκαν, πρέπει να πω ότι πάντα οι πρόεδροι έρχονται για να ακούσουν ε, επικρίσεις, αλλά όλοι αναγνωρίζουμε τελικά πόσο δύσκολη είναι η εργασία που επιτελείται. Στο τέλος λοιπόν ακούγονται και έπαινοι. Ξέρουμε ότι η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πήρατε το βάπτισμα του πυρός και όντως ανταποκρίνεστε σωστά και παίρνετε τις σωστές αποφάσεις. Στην, ε, θα φύγω, σε λίγο θα εγκατέλειψω την Προεδρία γιατί έχω να πάω σε μια άλλη συνεδρία. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους απλώς ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε τις ψηφοφορίες αλλά πρέπει να ορίσουμε και ένα μέλος που θα μας εκπροσωπήσει ε, στην ε, Συμβουλευτική Επιτροπή Στατιστικών. Εγώ ήμουν μέλος το 2008, γιατί μου εισηγήτρια τέτοιου θέματα, αλλά παρετήθηκα, δεδομένου ότι έχω το δύσκολο χρέος να προεδρεύω. Ο κύριος Σικλούνα είναι υποψήφιος για την θέση αυτή. Οι συντονιστές το αποφάσισαν και θα ψηφίσουμε επισήμως αυτό τον ορισμό σήμερα το απόγευμα και τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίες θα διαβιβαστούν στην διάσκεψη του πρόεδρου θα πάρουν τελική απόφαση. Αυτό ήταν ενημερωτικό λοιπόν για τις ψηφοφορίες σήμερα το απόγευμα. Ε, το λέγω για αυτούς οι οποίοι δεν ήταν παρόντες στην προηγούμενη θητεία. Τώρα θα ήθελα να δώσω την Προεδρία στον Έντουατ Συγκλούνα, τον ίδιο. για το υπόλοιπο πρωινό. Ευχαριστώ. Um, uh, Μπορούμε να συνεχίσουμε με, την επόμενη, με το επόμενο τμήμα της συνεδρίασης και πρωτού σας ε, παρουσιάσω τον κύριο Κωνσταντσίου. έχω μια σύντομη ανακοίνωση να σας κάνω. γίνει ανοιχτή συνεδρίαση συντονιστών με τον πρόεδρο του EFC, τον κύριο Τόμας Βάιζερ, την 3η ε, 8 Μαΐου μεταξύ 2 και 3 το απόγευμα. Το EFC παίζει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες ε, ελλείμματος που βρίσκονται σε εξέλιξη και έτσι θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να συζητήσουν τις εξέλιξεις στον τομέα αυτό συμπεριλαμβανομένου του χρονικού πλαισίου για την διόρθωση των υφιστάμενων ε, ελλημάτων. Πολύ ωραία. Και περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων τώρα με την... Ε, μετά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Βίτορ Κωνστανσίο. Η παρουσίαση έχει να κάνει με την ετήσια έκθεση, όπως προείπα, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ό,τι αφορά το προηγούμενο έτος. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά την νομισματική πολιτική και να επανέλθουμε σε θέματα δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά την τραπεζική συνεργασία, την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ε, τα λοιπά. Όλα αυτά, ε, μάλλον ο λόγος θα δοθεί σε διαδικασία Κάτσου the Οι συντονιστές θα κληθούν να κάνουν ερωτήσεις πρώτοι μετά την παρουσίαση. Κύριε Κωνσταντσίο, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Νομισματικών Οικονομικών Υποθέσεων, με μεγάλη ευχαρίστηση είμαι πάλι εδώ και θα σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2011, που είναι μέρος στις υποχρέωσεις που έχουμε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ σύντομα πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στις νομισματικές και οικονομικές εξελίξεις του τελευταίου χρόνου και θα αναφέρω ποιες είναι οι δικές μας αποφάσεις. Θα μιλήσω για τις ε, παρούσες δημοσιονομικές προκλήσεις στην Ευρωζώνη και την πρόοδο που επιτεύθηκε για την ενίσχυση του πλαισίου ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και θα σας αναφερθώ σε θέματα δημοσιονομικής σταθερότητας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω κάτι σημαντικό για το 2011 το γεγονός ότι έχουμε στην Ευρωζώνη ένα νέο 17ο μέλος στην Εστονία, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται πόσο σημαντικός ρόλο παίζει ε, στην διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης η Ευρωζώνη στην οποία συμμετέχουν χώρες και οικονομίες που πληρούν τα κριτήρια προσχώρησης. Το 2011 συνέχισε να είναι ένας ε, χρόνος στον οποίο συνέβησαν εξαιρετικά γεγονότα και αντιμετωπίσαμε συνθήκες ε, μεγάλης πρόκλησης σε θέματα οικονομικά και νομισματικά στην τράπεζα. Στις αρχές συνέχιζε να υπάρχει ε, οικονομική ανάκτηση στην περιοχή της Ευρωζώνης με γενικότερη ανάπτυξη, αύξηση της εσωτερικής ζήτησης, αλλά αυξήθηκε το ποσοστό πληθωρισμού στις αρχές του 2011 εξαιτίας της αύξησης της τιμής της ενεργειακής και των πρώτων υλών, πράγμα το οποίο οδήγησε σε αύξηση και του πληθωρισμού και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών, και να μειώσουμε την κερδοσκοπία σε θέματα πληθωριστικά, αποφασίσαμε να αυξήσουμε το βασικό ε, επιτόκιο τον Απρίλιο και τον Ιούλιο κάθε φορά κατά 0,25%. Δεδομένου ότι για δύο χρόνια είχαμε διατηρήσει το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Το μέσα του Ιουλίου ε, δημιουργήθηκαν διάφορες εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να ανακτηθεί στην ε, αγορές η εμπιστοσύνη, αποφασίσαμε να μειώσουμε ε, και να αποκτήσουμε την, συγγνώμη, την εμπιστοσύνη ε, δεδομένου ότι υπήρχε παγκοσμίως μείωση της ζήτησης, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε τις οικονομικές δραστηριότητες το δεύτερο εξάμεινο του 2011. Και οι μεγάλες αβεβαιότητες μαζί με την απομόχλευση και τις πιέσεις που δημιουργούνταν στους συλλογισμούς των τραπεζών ξέρουμε ότι δημιούργησαν προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, πράγμα το οποίο μας οδήγησε σε μείωση του βασικού επιτοκίου ε, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο συνολικά κατά 0,50%. Ε, δεδομένου ότι οι, χρηματοπιστω... οι εντάσεις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, ε, δημιούργησαν προβλήματα στη νομισματική πολιτική, αποφασίσαμε επίσης να υιοθετήσουμε μία σειρά μη, αν θέλετε, εκτάκτων νομισματικών μέτρων τον Αύγουστο του 2011, όπως το, το πρόγραμμα των ε, τίτλων και ε, χρεογράφων ε, το λανσάρισμα ενός δεύτερου προγράμματος καλυμμένων ομολόγων και μέτρα για να μπορέσουμε να παρέχουμε ρευστότητα σε ξένα νομίσματα. Επίσης, αποφάσισε το ευρωσύστημα να διατηρήσει τη διαδικασία σταθερών επιτοκίων ανακατανομής όσον αφορά τις ε, αναχρηματοδοτικές πράξεις. Το Δεκέμβριο, επίσης, υιοθετήσαμε διάφορα μέτρα για να υποστηρίξουμε τις πιστώσεις, τις πιστώσεις με, την, με διάφορες πράξεις αναχρηματοδότησης τριεστούς διάρκειας, με την αύξηση των εγγυήσεων και τη μείωση του επιτοκίου στο 1%. Αυτό για να μπορέσουμε να ε, βοηθήσουμε τον ε, ευρωτραπεζικό τομέα και να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις των περιορισμών που υφίστανται οι αγορές. Ε, η κρίση ε, απέδειξε ότι, ότι η διασφάλιση ε, υγιών κρατικών προϋπολογισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική ε, σταθερότητα. Ε, ως αποτέλεσμα, η ενοποίηση των, του γενικού ε, κρατικού A Ελλείμματος στην περιοχή της Ευρωζώνης έπεσε σημαντικά από 6,2% του ΑΕΠ το 2010 σε 4,1% του ΑΕΠ το 2011. Αυτή η μείωση του ελλείμματος προπολογισμού επιτεύθηκε μέσω της μέτρων εξυγίανσης και υποστηρικτικών μέτρων για να μπορέσουμε να ε, βοηθήσουμε τις κυκλικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά. Ένα κύριο χαρακτηριστικό ε, των αγοράς ε, χρεογράφων στις χώρες της Ευρωζώνης το 2011 ήταν η διαφοροποιημένη εξέλιξη των αποδόσεων στις διάφορες χώρες ως αποτέλεσμα της διαφορετικής ε, δημοσιονομικής πολιτικής κάθε Η δράση των κεντρικών τραπεζών είναι να υποστηρίζουν τη ρευστότητα του συστήματος και τελικά μπορώ να πω ότι μπορέσαμε να επιτύχουμε πρόοδο για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης ε, της ε, Ευρωζώνης για να προλάβουμε τις κρίσεις και για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Οι ε, κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πω ότι ενισχύθηκαν και καθώς και το νομικό πλαίσιο των διαφόρων κρατών μελών ενισχύθηκε ένα νέο μακροοικονομικό πλαίσιο εποπτείας δημιουργήθηκε και οι νέες διατάξεις ε, περιλαμβάνουν στοιχεία ε, σημαντικά για να προχωρήσουμε προς την ε, κατάλληλη διεύθυνση. Παρ' όλα αυτά πάντα ο διάβολο κρύβεται όπω λέμε στι λεπτομέρειε εφαρμογή και κυρίω το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2010 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει ο μηχανισμός επιτήρησης ε, να ενισχυθεί. Η τράπεζα θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο διαχείρισης της κλίσης μαζί με την Επιτροπή, το Διεθνές Νομικοτικό Τραμείο Διεθνέ Μεσογειακό Ταμείο θα αναλάβουμε τις διάφορες αναλύσεις των ε, των ε, κρατικού χρέους για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις χώρες μέρες που το χρειάζονται μέσω του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητες. Χαιρετίζουμε επίσης την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, το οποίο θέλει να αυξήσει ε, σε περίπου 800 δις ευρώ το ε, ποσό προστασίας για το ευρώ. Θα πρέπει παρόλα αυτά να είμαστε σαφείς, τίποτε δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει τις απαραίτητες ε, διαρθρωτικές και δημοσιονομικές προσαρμογές που πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Τώρα, α αρχίσω να ασχοληθώ με θέματα που αφορούν το χρημα, δημοσιονομικό τομέα. Θα αρχίσω με ό,τι αφορά τις τράπεζες, με την εισαγωγή του CRD. CRR, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η πρώτη που θα αρχίσει να εφαρμόζει τις συμφωνίες της Βασιλείας 3. Όπως προχωρούμε, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι υποστηρίζουμε την ε, θέσπιση ενός ενιαίου συνόλου ευρωπαϊκών κανόνων για, τις χρηματοπιστωτικές, για τα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα, ε, ώστε να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τους κανονισμούς διατησίας και τις τρευλώσεις της ανταγωνιστικότητας, ώστε να μπορέσουμε να θεσπίσουμε ε, απαιτήσει προσεκτικά όταν υπάρχει πρόβλεψης κινδύνου για το όλο σύστημα. Είναι λοιπόν σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια τα κράτη-μέλη να μπορέσουν προσωρινά να μειώσουν τα ε, ποσοτιαία ποσοστά και τις ε, πολιτικές που θα κάνουν ώστε να μην υπερβούν τα πλαίσια που ε, προβλέπονται από τους ορισμούς. Εμείς θέλουμε σε όλα αυτά τα μέσα που θα θεσπιστούν να συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό του κεφαλαίου, οι μεγάλες εκθέσεις, το ποσοστό ρευστότητας, το ποσοστό μόχλευσης έτσι όπως έχει ε, δημοσιευθεί και στην ε, αιτιολογημένη γνωμοδότηση που κάναμε. Το γεγονός ότι θα υπάρχει διαφορετικά μέτρα μακροπρόθεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, περιοχή της Ευρωζώνης, όπου η ενιαία νομισματική πολιτική που εστιάζεται στις, ε, ε, σε μέσους κοινού όρους δεν επιτρέπει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν νομισματικά μέτρα στα πλαίσια της πολιτικής που υιοθετούν για να μπορέσουν να αποφύγουν εκρήξεις των πιστώσεων και ε, έλλειψη ευθυγράμμισης των ε, τιμών που ισχύουν στις χώρες τους. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξουν ε, σε συμφωνία για όλα αυτά τα μέσα τα οποία θα παρουσιάσουμε στο μέσο, το καλοκαίρι αυτού του έτους. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, προβλεπόμενη μεταρρύθμιση του πλαισίου του κοινοτικού για τα χρεόγραφα και για τα παράγωγα στα πλαίσια των κανονισμών τα οποία προβλέπονται από το 2011. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη συμφωνία για τον κανονισμό ΕΜΙΡ και για το ε, που, θα που εφαρμόζει η εντολή του G20 για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την αντίσταση των ε, αγορών παραγόγων OTC. Συγχρόνως πρέπει να πω ότι χαιρετίζουμε την ε, αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα των αγορών και υποστηρίζουμε τον αντικειμενικό στόχο ε, που περιλαμβάνεται ε, στην πρόθεση Επιτροπής για τους οίκους ε, πιστοληπτικής ικανότητας. Θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από αυτούς και το ίδιο το ευρωσύστημα ε, δεν θα πρέπει μηχανικά να εξαρτάται μόνο από αυτού του είδους τις αξιολογήσεις, δεδομένου ότι σε κάθε μέθοδο που ακολουθείτε υπάρχουν περιορισμοί. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την χρησιμοποίηση του πλαισίου εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλες αυτές οι κανονιστικές ε, ε, πρωτοβουλίες που προβλέπονται για την ενίσχυση της ενίας νομισματικής αγοράς και των υποδομών θα συμπληρωθούν από το, ε, το, το πάρα πολύ σημαντικό έργο που είναι το Target to Securities που προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το 2015. Έχουμε αρχίσει εδώ και δύο χρόνια περίπου, μετά από δύο χρόνια συγγνώμη, ε, διαπραγματεύσεων, έχουμε με τα CDS, με τα CSDs, έχουμε την πεποίθηση ότι το σύστημα θα μπορέσει να λειτουργήσει ε, σύντομα. Τώρα, θα ήθελα να αφαιρθώ στην διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων. Υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εισαγάγει ένα νέο πλαίσιο για την ανάκτηση των τραπεζών και την ε, επίλυση των προβλημάτων για να μπορέσουμε να ε, αντισταθμίσουμε τα παρόντα εμπόδια που υπάρχουν για την διαχείριση κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να οπλιστεί με μία σειρά μέτρων όπως σχέδια ε, ανάκτησης και διευθέτησης των προβλημάτων, διαχωρισμό του ενεργητικού και να μπορέσει ε, να ανταποκριθεί στα σημερινά προβλήματα. Αναφέρομαι ιδιαιτέρως ε, στην συμβολή του ιδιωτικού τομέα, στα περίφημα PCI, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν χωρίς να δημιουργηθούν αντίστροφα αρνητικά αποτελέσματα στην χρηματοδότηση των τραπεζών. Και ε, ίσως θα πρέπει οποιοδήποτε απόφαση για την χρησιμοποίηση των ε, PCIs να καθυστερήσει για κάποια χρόνια. Παρ' όλα αυτά ε, πρέπει να πω ότι οποιαδήποτε ε, συμμετοχή υποχρεωτική του PCI του ιδιωτικού τομέα ε, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Ε, ξέρουμε ότι τα μικρότερα πιστοτικά ιδρύματα δεν μπορούν με ευκολία να διοχετεύουν στην αγορά τέτοιου είδους χρεόγραφα προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Ε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό για την επίλυση των προβλημάτων αναφέρουμε στην, είναι η δημιουργία του Ταμείου Εξυγίανσης το οποίο θα, μπορούσε να, θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και να παίξει σημαντικό ρόλο κυρίως για την ε, διευθέτηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα διασυνοριακά τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, ενδεχόμενα προβλέπεται να δημιουργηθεί αργότερα ένα ευρωπαϊκό ταμείο των ταμείων εξυγίανσης αν θέλετε για να μπορέσουν να επιληθούν όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα. Δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ε, όσον αφορά το καθεστώ που θα επικρατήσει για τις πλήρη διαφάνεια, πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι προτάσει Ευρωπαϊκής Επιτροπή να γίνουν γνωστές πριν από το καλοκαίρι. Τελικά επιτρέψτε μου να πω ε, κάποια λόγια για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ε, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να μπορέσει να αυξηθεί η αντίσταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα σε σχέση με την γενικότερη χαλάρωση που επικρατεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ε, ξέρουμε ποιες είναι οι προτάσεις τις οποίες κάνει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και ξέρουμε ότι θα πρέπει να ε, μπορέσει να ανταποκριθεί στα προβλήματα της οικονομίας σήμερα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πάρα πολύ ισχυροί. Κυρίες και κύριοι, το 2011 Αναμφίβολα ήταν μια χρονιά προκλήσεων για την Ευρωζώνη, κυρίως ε, εξαιτία των τρομερών προβλημάτων που δημιουργήθηκε στο δημόσιο χρέος ε, κάποιων χωρών και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχω εμπιστοσύνη στα προγράμματα οικονομικής διακυβέρνησης και στις μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν και ως συν νομοθέτης η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζω ότι θα μπορέσει με τους κανόνες που θα υιοθετήσει να συνεισφέρει στην αύξηση της σταθερότητας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κωνστανσιο. Να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Νομίζω πρώτος, πρώτη είναι η Σιλβί Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας. Δεν είμαστε πολλοί, αλλά είναι σημαντικό παρόλα αυτά. Θα ήθελα να αναφέρω δύο σημεία από τα πολλά πράγματα που είπατε στην παρουσίαση σας. Το πρώτο, με τον κύριο Ντράγκη, μιλήσαμε γι' αυτό. Εγώ ήθελα να κάνω έκκληση για να γίνει πιο διαφανής η ανακοίνωση. Όχι να δημοσιεύσετε τα πρακτικά και όλα αυτά, αλλά όσον αφορά τις μη συμβατικές ε, πράξεις. Πιστεύω είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί κατάλληλα, πιστεύω, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να εξηγήσουμε και στους ε, πολίτες που πήγαν τα χρήματα. Η απάντηση που μας έδωσε ο κύριος Δράγκη, που την καταλαβαίνω, που μας λέει ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα πριν επανέλθουν τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν δημιουργήσει τα χρήματα ρευστότητα στο σύστημα, έχουν περάσει από το ένα μέρος στο άλλο εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά θα ήθελα, αν μπορείτε να προσπαθήσετε, δεν ξέρω πώς θα ήταν δυνατόν, να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία, ώστε να είναι πιο σαφές, ε, ε, να άρουμε αυτό το πέπλο μυστηρίου από το τι συμβάνει. Εδώ μιλάμε για ένα τρισεκατομμύριο, είναι τεράστιο ποσό, πιστεύω σε ένα... Ε, σύστημα δημοκρατικό. Θα πρέπει να μπορούμε να υπάρχει εχνηλασιμότητα, να ανοιχνεύσουμε πού είναι τα χρήματα. Το κάνουμε και για τι Αγελάδε. Δεν το λέω επικριτικά. Ε, να, να απομυθοποιήσουμε κάποιες ε, ε, επικρίσεις που ακούγονται. Είχαμε μια εκστρατεία κατά της Ευρωπαϊκής και της Κεντρικής Τράπεζας στη Γαλλία. Εγώ προσπάθησα να επαναφέρω τα πράγματα σε μια σωστή ισορροπία. Η έκθεσή σας είναι ιδιαίτερα πλήρης, απλά ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε αυτό το σημείο. Εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε τη μάχη της επικοινωνίας, θα την κερδίσουν οι ακραίοι. Το δεύτερο που ήθελα να πω εγώ ήμουν εισηγήτρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Συστημικό Κίνδυνο, για τη δράση αυτού, αυτής της Επιτροπής. Πρόκειται για ένα νέο όργανο που μόλις ξεκινάει. Εγώ επαναλαμβάνω εδώ αυτό που είπα πολλές φορές και στην Οβλομέλεια και στον κύριο Ντράγκη. Μας απασχολεί η διατήρηση της ενιαίας αγοράς. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε, το Single Rule Book να είναι ένα πραγματικό βιβλίο ενιαίο βιβλίο κανόνων. Μπορούμε να φανταστούμε ότι υπό ιδιαίτερε περιστάσεις μπορούμε να έχουμε κάποιο περιθώριο ευελιξία. Αλλά εάν δεσμευτούμε όπως φαίνεται να θέλουμε να κάνουμε με σε ενό είδου εξουσιοδοτήσεις που δίνονται στους εθνικούς νομοθέτες, όχι επίπεδο 2, στο αρχικό επίπεδο, πιστεύω ότι εδώ αποδομούμε αυτό που έγινε με μεγάλο κόπο ο Ζακ Ντελαροζιέρ είχε ε, ε, συζητήσει με τον Τζακ Ροζιέρ που ήταν πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Η έκθεση Ντελαροζιέρ προέβλεπε ένα περιθώριο ευελιξίας αλλά όχι την αμφισβήτηση της αρχής του single book. Είναι καλό αυτό διότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας δύσκολης κρίσης και πρέπει να αντέξουμε. Έχουμε τις εθνικιστικές ιδέες που επανέρχονται και πρέπει να τις αποθήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να σας δώσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας κύριε Αγκουλάου. Για την πρώτη αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι απόλυτα όσα λέτε, αλλά κατά, από πολλές απόψεις ε, αυτό που ζητάτε ουσιαστικά με την εγκλήση σας είναι αδύνατο. Ένα από τα χαρακτηριστικά του χρήματος είναι ότι τα χρήματα κινούνται. Δημιουργούνται, μπαίνουν σε κίνηση και μετά θεωρητικά είναι αδύνατον ουσιαστικά πραγματικά να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πού ακριβώς πήγαν συγκεκριμένα ποσά. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα LTRO αύξησαν τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Όχι κατά ένα τρισεκατομμύριο, όπως λέγεται συνήθως, αλλά μόνο κατά μισό τρισεκατομμύριο. Γιατί, διότι άλλες μορφές χρηματοδότησης των τραπεζών μειώθηκαν. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν λιγότερο άλλους μηχανισμούς ώστε να αξιοποιήσουν τα LTRO μακροπρόθεσμα. Η αύξηση αυτή ήταν μόνο εισαγωγικών μισό τρισεκατομμύριο. Αυτό λοιπόν είναι σημαντική πληροφορία ήδη. Διότι μας παρουσιάζουν λανθασμένα το όλο ποσό. Τι συμβαίνει στη συνέχεια. Πιστεύω ότι όντω πρέπει να εξηγήσουμε περισσότερα, παρότι εδώ μιλάμε για τεχνικέ λεπτομέρειε όσον αφορά τη δημιουργία των χρημάτων και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, ορισμένοι άνθρωποι είναι προβληματισμένοι. Δεν καταλαβαίνουν πώ εμεί παρέχουμε τέτοια ρευστότητα, ενώ ταυτόχρονα σχεδόν το ίδιο ποσό υπάρχει σε καταθέσει των τραπεζών. Σε εμά. Συνολικά αυτό είναι μια ανάγκη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αυξής, αυξάνοντας την μονομισματική βάση αυτή αυξάνεται εάν οι τράπεζες επαναπληρώσουν αυτές τις συμφωνίες επαναγοράς μετά από ένα ή από τρία έτη ή αν θα πουλήσουμε ενεργετικά από το ισοζύγιο μας ε, διαφορετικά η, η αύξηση παραμένει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά παραμένουν ακίνητα και δεν φέρουν αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν σε τεράστιο βαθμό μεταξύ των τραπεζών του συστήματος. Όπως είπαμε ήδη, δημοσίως οι τράπεζες που δανείστηκαν περισσότερο με αυτές τις δύο δράσεις δεν είναι πλέον καθόλου οι τράπεζες που έχουν τις πιο μεγάλες καταθέσεις σε εμάς. Δεν είναι οι ίδιες τράπεζες δεν είναι καν οι ίδιοι τραπεζικοί τομείς. Τα χρήματα κυκλοφόρησαν σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και φυσικά χρηματοδοτούν τα ισοζύγια των τραπεζών. Κάτι άλλο που δεν αναφέρεται επαρκώς και το έχουμε εξηγήσει. Μία από τις αιτίε που προέβημεν σε αυτές τις δράσεις ήταν επειδή οι τράπεζες το πρώτο τρίμηνο του 2012 αντιμετώπιζαν επαναχρηματοδότηση τραπεζικών ομολόγων που είχαν φτάσει σε ορίμανση και έπρεπε να τα εξοφλήσουν σε ύψος 230 δισεκατομμυρίων και η αγορά έκδοσης τραπεζικών ομολόγων είχε κλείσει στο τελευταίο μέρος του περασμένου έτους. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν μεγάλο μέρος της ρευστότητας που παρήχαμε από τις τράπεζες για την εξόφληση των ε, οριμασμένων ομολόγων επειδή δεν μπορούσαν να εκδώσουν στην αγορά τα ίδια ομόλογα για να εξοφλήσουν τα προηγούμενα. Ένα πολύ λοιπόν μεγάλο κομμάτι της ρευστότητας που παρήχαμε χρησιμοποιήθηκε από τις τράπεζες για την εξόφληση χρέους που είχαν και που είχε φτάσει σε ορίμανση στο πρώτο μέρος του έτους. Αυτό είναι για να σας δώσω απλά ένα παράδειγμα. Αλλά όπω σας είπα τα χρήματα κινούνται για να αποκτήσετε μια εικόνα. Το συνολικό ισοζύγιο των πληρωμών στην Ευρωζώνη ανέρχεται σε 32,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές καταθέσεις στις τράπεζες, στο σύνολό τους, ανέρχονται σε 20,4 εκατομμύρια. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσετε μια εικόνα της κλίμακας των επιπλέον 500 δισεκατομμυρίων ρευστότητας που παρήχαμε στις τράπεζες και που ουσιαστικά μπήκαν στο σύστημα σε όλες τις χώρες κινήθηκαν μέσα στο σύστημα όλων των χωρών διότι όπως είπε ο Πρόεδρος πριν από λίγο από τις 800 τράπεζες που συμμετείχαν στο δεύτερο LTRO ένα μεγάλο κομμάτι ήταν από τη Γερμανία Καταλαβαίνετε λοιπόν την πολυπλοκότητα αυτής της διαδικασίας δημιουργίας χρήματος Αυτά τα στοιχεία, ωστόσο, που σας αναφέρω εγώ αυτή τη στιγμή, τα έχουμε ήδη εξηγήσει, αλλά συμφωνώ μαζί σας, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και να εξηγούμε καλύτερα στο κοινό τι σημαίνουν όλα αυτά. Διότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι, οι πολίτες να καταλάβουν. Και ακούω ερωτήσεις και εδώ, οι οποίες δείχνουν ότι, ότι δεν κατέχουν όσοι ρωτούν τις, τις λεπτομέρειες της δημιουργίας χρήματος. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας πιο σύντομα, για ποιο πράγμα κάνουμε έκκληση. Κάνουμε έκκληση ώστε σε προσωρινή βάση, προσωρινή, εάν σε μια συγκεκριμένη χώρα της Ευρωζώνης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρξει credit boom, πιστοτική φούσκα ουσιαστικά ή ε, φούσκα ακινήτων και ειδικότερα εντός της Ευρωζώνης. Δεν έχουμε εθνική νομισματική πολιτική. Ποιοι μηχανισμοί λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εν λόγω χώρα για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος που όπως είδαμε σε ορισμένες χώρες δημιούργησε σημαντικότατα προβλήματα. Οι μόνοι μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν θα είναι προσωρινά ενώ υπάρχουν αυτές οι συνθήκες να αυξήσουν, να ενισχύσουν ορισμένους από τους μηχανισμούς μακροοικονομικής πολιτικής. Αυτό λοιπόν υπάρχει διαθέσιμο. Κατά την άποψή μας όμως, αντίθετα με κάποιους άλλους, δεν μπορεί να γίνεται μόνιμη χρήση αυτών των μηχανισμών. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε gold plate banks όπως λέμε στην τράπεζα με υψηλότερα κεφάλαια όπως υπάρχουν σε ορισμένες χώρες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι προσωρινή χρήση αυτών των μηχανισμών όταν υπάρχουν λόγοι που αιτιολογούν τη χρήση αυτών των μηχανισμών. Και πάντα υπό δύο προϋποθέσεις μόνο για την ενίσχυση και όχι την αποδυνάμωση και χωρίς αλλαγή των ορισμών. Διότι σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθεί χάος και θα καταστραφεί το single rule book. Απλά να αλλάξει η ε, εξισορρόπηση κατά κάποιο τρόπο. Αυτή είναι η θέση μας και εμείς κάνουμε έκκληση να θεωρήσετε ότι αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία της, Ευρωπαϊκής, της Νομισματικής Ένωσης. Ευχαριστώ. Έχουμε τρεις ομιλητές. Τον Διέγκο κυρία Άννη Ποδημάτα. Διέγκο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Κωνστάνσιο. Θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ θετική η παρουσίαση που κάνατε, διότι αναφερθήκατε στην έκθεσή σας στην σταθερότητα και στην εμπιστοσύνη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Και δίνω ως παράδειγμα αυτά τα οποία συνέβησαν πέρσι με την, ε, τον πληθωρισμό. Η κυρία Σιλβί Γκουλάρ έθεσε ένα θέμα σχετικά αφορά την επικοινωνία. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εάν ε, θέλετε είναι στο στόχαστρο όλων. Με μεγάλη προσοχή όλοι παρακολουθούν τι θα πείτε, εσείς και ο διευθυντής σας. Άρα ο ίδιος ο ρόλος σας ε, αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικός και δημιουργείται προσδοκίες. Και όπως ξέρουμε κάποια από αυτά που λέτε πολλές φορές ε, την χάνουν διαφορετικής ερμηνείας. Στην ε, ε, Πορτογαλία πριν ε, από 15 μέρες ελέγχθη κάτι για την ε, θέση της Πορτογαλίας στις ευρωπαϊκές αγορές, αρνητικό, αλλά μετά από 15 μέρες ελέγχθη ότι όντως τώρα επιστρέφει η Πορτογαλία στις ευρωπαϊκές αγορές, πράγμα το οποίο δημιούργησε εμπιστοσύνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό το οποίο είναι σημαντικό για τα άτομα είναι πώς βλέπει τα πράγματα σε σχέση με τις προσδοκίες που υπάρχουν. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρου όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης. Είπαμε ότι σε κάποιες χώρες όπως ε, στην Ιρλανδία όπως και στην Πορτογαλία θα πρέπει σε ε, συνεργασία με την Τρόικα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα διάφορα προγράμματα ε, για την βελτίωση των ε, οικονομιών μας. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη λιτότητα, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η περίφημη ανάπτυξη την οποία θέλουμε και ε, πολλοί γνωρίζουν ότι τα μέτρα λιτότητας θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα αλλά δεν να τα επιλύσουν. Το 2011 μπορεί να δοθεί σαν καλό παράδειγμα του που οδήγησε το πρόγραμμα λιτότητος που εφαρμόστηκε. Και πολλές φορές, και τώρα ξεπερνώ λίγο τα πλαίσια της παρουσίασής σας, πολλοί λέγουν ότι σήμερα ζούμε την κρίση που ζούμε δεδομένου ότι δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε σωστά την πολιτική που χρειαζόμαστε με το ευρώ. Γι' αυτό προβλέφτηκε αυτό το six pack για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε και θα πρέπει επίσης να δούμε σήμερα πώς θα μπορέσουμε να χειριστούμε ε, την αγορά των τίτλων και χρεογράφων στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Και τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Ε, μου επιτρέπετε, θα απαντήσω κι εγώ στα πορτογαλικά, στη γλώσσα μου. Στο σύνολο των ερωτήσεων που έκανε ο συναδελφός σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ότι θεωρείτε θετικά αυτά τα οποία είπα για την έκθεσή μας. Τώρα, το θέμα της ε, επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικό, αλλά πολύ δύσκολο όπως ξέρετε. Ένα από τα παραδείγματα που δώσατε, δηλαδή αν ακούσει κανείς ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία είπα, μπορεί να δημιουργηθεί ε, μια αρνητική ε, εντύπωση για την ε, Πορτογαλία. Εγώ ποτέ μου δεν είπα σφαιρικά ότι θα μπορούσε να έχει πρόβλημα τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, διότι το σενάριο στο οποίο εμείς δουλεύουμε και με το οποίο συνεργαζόμαστε και με την Τρόικα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μέτρα για να βελτιώσουμε την κατάσταση χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι δίνουμε εγγύηση 100% ή δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέρος. Αλλά αυτό είναι το σενάριο το οποίο ακολουθούμε βάσει πραγματικών γεγονότων. Το γενικότερο πρόβλημα της ε, εξυγίανσης το ανέφερε ο πρόεδρος Δράγκη την προβληματική όλων των κρατών, στα, διότι υπάρχουν κράτη που δεν έχουν καμία άλλη δυνατότητα παρά να αντιδράσουν στις πιέσεις των αγορών και να μειώσουν το δημόσιο έλλειμμα τους και είναι όντως αληθές ότι με εξωπρόθεσμα δεν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των συνθήκων που απαιτούνται για να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Αλλά το έχουμε πει, το είπε και ο πρόεδρος Δράγκη πολλές φορές και εγώ ο ίδιος ότι βράχει πρόθεσμα είναι προφανές ότι οι συνθήκες ε, οι παρούσες και τα προβλήματα των ε, ε, κρατικών προϋπολογισμών δημιουργούν πρόβλημα για την ανάπτυξη. Βραχυπρόθεσμα λέγω. Θα πρέπει λοιπόν να ξανατεθούν οι όροι για μια ε, αυξημένη οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Κοιτάξτε τώρα, τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη συνολικά. Το 2011 σας είπα ότι μειώθηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού γενικότερα. Σε σχέση τώρα με το τελευταίο μέρος της ερώτησής σας για τις μεταρρυθμίσεις, οι μεταρρυθμίσεις όπως είπατε, τι σημαίνει. Τι σημαίνουν ότι κάποια θέματα της οικοδόμησης της ΟΝΕ καταρχάς οι ευθύ εξ αρχής μάλλον δεν ελήφθησαν υπόψη. Ποια είναι τα διδάγματα τα οποία πρέπει να συνάγουμε από όλη αυτή την κρίση την οποία διέρχεται η Ευρωζώνη. Πρώτα απ' όλα, ότι η ΟΝΕ απαιτεί μεγαλύτερη ε, ενότητα, αν θέλετε, για την πολιτική προπολογισμού από κάθε χρόνο. Θα πρέπει δηλαδή να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις που πήραμε κυρίως πρόσφατα. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί αντιμετώπισης των κρίσεων. Πράγμα το οποίο δεν είχε προβλεφθεί ευθύ εξ αρχή. Όταν δημιουργήθηκε η ΟΝΕ, είπαμε ότι όντω θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει μία νομισματική κρίση, αλλά όχι με τις σημερινές της διαστάσεις. Και κάτι που μάθαμε επίσης από την κρίση είναι ότι μάθαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένωση χρηματοπιστωτική. Οι συνθήκες λοιπόν εποπτείας και επίλυσης των κρίσεων του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει αν θέλετε, όπως είπα και στην παρέμβασή μου, να έχουν πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Πρόκειται λοιπόν για τρία μαθήματα που μάθαμε από την κρίση και αυτό που μάθαμε θα πρέπει να το εφαρμόσουμε κάνοντας τις απαραίτητες αναπροσαρμογές για να διορθώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η Άννη Ποδηματά. Uh, σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, τέννη σας παρουσίαση, στην οποία σωστά υπογραμμίσατε εκ νέου τη σημασία να πετύχουμε χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Νομίζω, κυρία Αντιπρόεδρε, ότι σε ό,τι αφορά την ανάγκη να διδαχτούμε από τα παθήματα και τις αιτίες που οδήγησαν στην τρέχουσα κρίση, νομίζω ότι είναι επιτακτικό να υπάρχει και το πολιτικό θάρρος για να αξιολογηθεί σωστά οι πολιτικές ε, και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία τρία χρόνια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Και νομίζω ότι μεταξύ αυτών των διδαγμάτων που θα πρέπει να εξαγάγουμε και μετά από αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, ο κύριος Φέγιο και ο Κιλάρ, Νομίζω λοιπόν ότι ένα από τα διδάγματα που θα πρέπει να εξαγάγουμε είναι ότι η δημοσιονομική πειθαρχία είναι απαραίτητη, δεν επαρκεί όμως αυτή για να δημιουργήσει τους όρους εκείνους που θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την υφιστάμενη κρίση. Ασφαλώς γνωρίζω ότι θα τονίσετε την ανάγκη να προωθηθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και πάλι σε περιπτώσεις και περιόδους κρίσης και ύφησης, καλές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά να αποφεύγουμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να βαθύνουν την ύφεση. Ο σκοπός μας είναι να την ξεπεράσουμε και αναφέρομαι στον αντίκτυπο που είχε η απόφαση στη χώρα μου την Ελλάδα, η απόφαση μείωσης των ε, ελάχιστων των κατατών μισθών στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίκτυπος ήταν όντως ε, περαιτέρω βάθυνση, όξυνση της ύφεση, χωρίς καθόλου να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Πέρα από την Ελλάδα όμως, κύριε Πρόεδρε, Επανέρχομαι στο σημείο του πόσο απαραίτητε ε, είναι η μακροοικονομική και η δομοσυνομική σταθερότητα. Θα συμφωνείτε ότι η μακροοικονομική και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν έχουν να κάνουν μόνο με συγκεκριμένους δείκτες, αλλά και με τις κοινωνικές συνθήκες, με τους κοινωνικούς όρους που υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Η κυρία Γκουλάρ μίλησε για την ε, άνοδο του εξτρεμισμού όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κοινωνικής ε, αστάθειας. Άρα, αυτή η κοινωνική κατάσταση, αυτή η κοινωνική όρη, οι κοινωνικές συνθήκες έχουν λεφτεί σοβαρά υπόψη ως τώρα ή μήπω έχουν κάπως υποτιμηθεί. Σας ανοσοχή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό το συγκεκριμένο σημείο και άλλες δύο ερωτήσεις, κύριε Αντιπρόεδρε, σε ό,τι αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη θέση σας, το είπατε και εσείς, το είπαν και οι συναδελφοί μου. Υπάρχουν ε, νέοι αυστηροί κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης, ένα καινούργιο δημοσιονομικό σύμφωνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν ε, συντρέχουν οι όροι για να, για να ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία σταδιακά θα οδηγήσει στην κοινή διαμόρφωση του χρέους στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη. Γιατί αυτό είπε και ο Πρόεδρος κ. Μπαρόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μήπως έχει έρθει η στιγμή να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση σε ό,τι αφορά την ανάγκη παράτασης ε, της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε συνδυασμό με τους νέους αυτούς κανόνες που έχουν εφαρμοστεί για την ε, δημοσιονομική πειθαρχία και για την, ε, τα μέτρα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας που αποτυπώνουν τις ανησυχίες κατανοητές και προφανείς ανησυχίες. Θα ήθελα εκ να σας υπογραμμίσω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε δύο πράγματα που βρίσκονται στο υπόβαθρο όλων των αλλαγών αυτών. Καταρχάς ότι η χρηματοπιστωτική κρίση στον κόσμο ήταν τεράστια και όλος ο κόσμος δεν έχει ακόμα ανακάμψει πλήρως. Η ανάπτυξη είναι αργή παντού. Η ιστορία μας διδάσκει ότι αν σε περίπτωση τέτοιας κρίσης ακολουθεί φυσιολογικά επί σειρά ετών μία περίοδος χαμηλής ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν είναι προκαθορισμένο κατά κάποιο τρόπο. Η Αμερικανική οικονομία, μάλλον ο κύριος Ρόντρικ, είπε ότι τα πρώτα δέκα χρόνια της Οικονομικής Ένωσης ήταν πάρα πολύ καλά και μετά τα πρώτα δέκα χρόνια και πάλι θα πήγαιναν τα πράγματα καλά αν δεν είχε παρουσιαστεί η οικονομική κρίση. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να, να έχουμε υπόψη. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι επί σειρά ετών κάποιες χώρες ανέπτυξαν τεράστιες ανισορροπίες και όταν ε, ήρθε η κρίση επικεντρώθηκαν οι αγορές ε, σε αυτές τις ανισορροπίες. Πριν ήταν ε, απεριόριστη σχεδόν η χρηματοδότηση των χωρών αυτών, χωρί να αναλογίζονται οι αγορέ του κινδύνου. Και ξαφνικά μπήκε φρένο στι ροέ προ τι χώρε αυτέ. Και αυτό είναι ένα γεγονό. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε τρόπο να αντικαταστήσουμε όλε αυτέ τι εισρωές προ τι χώρε αυτέ. Οι χώρε αυτέ θα πρέπει να προσαρμοστούν, θα πρέπει να μειώσουν τι ανασορροπίες. Αυτό είναι το υπόβαθρο το οποίο πολύ καλά γνωρίζετε ασφαλώ και το οποίο και αναφέρατε άλλωστε. Δεν σα ε, διορθώνω. Απλά τονίζω κάποια στοιχεία, δύο στοιχεία που θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη για να μπορούμε να ακτιμούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα κοινωνικά προβλήματα. Ναι, ανάπτυξη σε κάποια τμήματα της Νομισματικής Ένωσης είναι αρνητική και θα συνεχίσει να είναι αργή για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό που θα πρέπει να εξηγήσουμε στις δημοκρατίες μας στους λαούς, στον κόσμο, είναι γιατί συμβαίνει αυτό και κάποιες από τις ε, ψευδεσίσεις που δημιουργούνται σε τέτοιες καταστάσεις νομίζω θα αντιγούσαν σε χειρότερα αποτελέσματα. Και τελικά όλα έχουν να κάνουν με τις λεπτομέρειες. Σε κάποια ζητήματα μπορούν να συζητηθούν, όχι η γενικότερη κατεύθυνση, αλλά τα επίπεδα μπορούν πάντα να συζητηθούν και θα πρέπει να συζητηθούν σε, με συγκεκριμένα παραδείγματα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει καμία γενική απάντηση. Να μην ξεχνάμε ότι εμείς ε, οι χώρες θα πρέπει να πείσουμε τις αγορές. για τη τελική ανάλυση με τις ανισορροπίες που υπάρχουν και τις αστάθειες οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν το χρέος τους, το χρέος των χωρών. Αν δεν γίνει αυτό, δεν υπάρχει 100% υποκατάστατο διαθέσιμο. Και αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις αγορές. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ποιες είναι οι αποφάσεις των αγορών και των επενδυτών. Τέλος. Τέλος, για τα δύο τελευταία ερωτήματα που θέσατε για την κοινή διαμόρφωση και ανάληψη του χρέους και για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την κοινή ανάληψη του χρέους. Προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατόν, θα έλεγα ότι θα χρειά... χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ε, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών, των κρατών μελών. Φυσικά τα μέτρα που λαμβάνονται τώρα προκειμένου να εμβαθυνθεί και η εποπτεία, η παρακολούθηση της ε, χρηματοοικονομικής κατάστασης ασφαλώς και θα ε, δυναμώσει, θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη εν αυτό χρόνο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της ευριονικής ε, ε, χρηματοοικονομικής ένωσης που ξεκινάει τώρα, αυτό θα το αποδείξει το μέλλον σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν μια διαρκής, ε, αέναη διαδικασία και θα συνεχίσει να είναι, θεωρώ, για την εντολή τώρα της τράπεζας. Ε, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Είναι πολιτική απόφαση των κρατών μελών. Εγώ απλά θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο, η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών είναι βασική, ουσιώδης για να δημιουργηθούν οι όροι για την οικονομική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εναλλακτική λύση στο σημείο αυτό και θα έλεγα ότι μέσω και μακροπρόθεσμα υπάρχει τεράστια συνένεση μεταξύ των όλων των σχολών οικονομολόγων. Γιατί Ιδάλως, όλες οι χώρες οι οποίες ε, επί αιώνες, επί δεκαετίες δημιουργούσαν πιο πολλά χρήματα, πιο πολύ πληθωρισμό, ήταν πιο ανεπτυγμένες. Δεν ισχύει όμως αυτό. Άρα η διασφάλιση σταθερότητας τιμών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Και αυτό δικαιολογεί την θητεία μας. Διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Και αυτή με τη σειρά της ε, θα διασφαλίσει άλλους στόχους, όπως και έχουμε ήδη πράξει. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Αν θέλεις να κάνεις ε, μια συμπληρωματική ερώτηση, δεν μιλάω για μια εναλλακτική. Μιλάω για μια συμπληρωματική σταθερότητα τιμών μίλησα για την παράταση της θητείας και της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όχι για την αλλαγή της θητείας και της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Λίαμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Υιοθετώντα το 2010 μέτρα όπως το S&P, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξοπλίστηκε με σημαντικά μέσα για να παρέμβει στους δευτερεύοντες αγορές του χρέους και έτσι βοήθησε να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία. Το 2011 η συνέχιση αυτών των μέτρων βοήθησε στην εγκαθίδρυση λίγο περισσότερο για τις αγορές και τους πολίτες στην ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ρεαλιστική, αντιδρά και είναι αποτελεσματική όπως είναι η Fed ή η Τράπεζα της Αγγλίας. Χρειαζόμαστε αυτόν τον παρεμβατισμό βασισμένο σε ρεαλισμό, ενώ η Ευρωζώνη ξαναμπαίνει σε ύφαση και αυξάνεται η ανεργία. Είναι απαραίτητο να αλαφρύνουμε τις μακροοικονομικές συνθήκες για να ευνοήσουμε την επιστροφή στην ανάπτυξη. Εμείς θεωρούμε ότι η νομισματική πολιτική από είναι ανεπαρκής. Γι' αυτό το λόγο οι Γάλλοι σοσιαλιστές θα ξανανοίξουν το, η συζήτηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Αλλά θα επανέλθουμε στην νομισματική πολιτική και τις προϋποθέσεις παρέμβασής της. Από αυτή την άποψη, πολύ συγκεκριμένες επιλογές έχουν γίνει. Ξεκίνησε το τέλος του 2011 ένα πρόγραμμα άνευ προηγουμένου για την επαναχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών τραπεζών εις βάρος μια πιο ισχυρή δράση για τα κρατικά χρέη. Μιλάω για τα LTRO. Το LTRO του, το έκτακτο του Δεκεμβρίου επέτρεψε την επαναχρηματοδότηση με ένα τρισεκατομμύριο με πολύ ευνοϊκές συνθήκες για τις τράπεζες. Ωστόσο, η κίνηση αυτού του προγράμματος ε, έγινε παράλληλα με την ε, μη χρήση πλέον του SMP που βοηθούσε στην επιστροφή σε μια σταθερότητα. Έτσι λοιπόν δεν έγινε καμία δράση εξαγοράς ε, κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ από τον Ιανουάριο του 2012. Αυτός ο επαναπρασανατολισμός ε, εις βάρος υπέρ των τραπεζών και κατά των κρατών είχε δυσάρεστες επιπτώσεις ε, παρότι τα επιτόκια στην Ισπανία για τα δεκαετία ομόλογα έπεσαν σε λιγότερο από 5% το Δεκέμβριο, ξανανέβηκαν και σήμερα υπερβαίνουν το 6%. Η εξέλιξη των Ιταλικών ομολόγων είναι παρόμοια. Δηλώσατε, κύριε Αντιπρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα ότι όταν ξεκινήσετε το πρώτο LTRO το Δεκέμβριο του 2011 δεν σας και πέρασε από το μυαλό ότι αυτό το πρόγραμμα θα έλυνε το, πρόγραμμα, το πρόβλημα του κρατικού χρέους. Το παραδέχεστε μαζί με εμά ότι σήμερα η προτεραιότητα δεν είναι να διασφαλίσουμε τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος που είναι ικανοποιητική, αλλά να καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία μεταξύ των κρατών κατά των κρατών μάλλον, που εμποδίζει τη δημοσιονομική εξυγίανση, ενώ κυκλοφορούν φήμες όλο και περισσότερο αγορές για τρίτο LTRO. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι αν συνεχίσει να υποβαθμίζεται η κατάσταση, η ΕΚΤ θα επιλέξει και πάλι ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα, όπως ε, έκανε επιτυχημένα από το 2010, ξανά ξεκινώντας το S&P. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο πρόεδρος Ντράγκη το ανέφερε. Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για μελλοντικά μέτρα. Μπορώ λοιπόν να απαντήσω στην τελευταία σας ερώτηση. Δεν μπορώ να απαντήσω στην τελευταία σας ερώτηση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το πρόγραμμα υπάρχει. δεν έχει διαγραφεί, δεν έχει καταργηθεί, υπάρχει. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ούτως ή άλλως, εάν συγκρίνεται με τις συνθήκες που υπήρχαν σε αυτό το τμήμα της αγοράς και στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής ε, τον Οκτώβριο, τότε τα πράγματα ήταν χειρότερα από τη σήμερα. Ακόμη και μετά από τις αλλαγές που προκλήθηκαν από τα προβλήματα επικοινωνίας της Ισπανίας, διότι ουσιαστικά τα σοβαρά προβλήματα της Ισπανίας προκάλεσαν την υποβάθμιση, την επιδείνωση της κατάστασης ε, και της τιμής του ισπανικού χρέους. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχουν μειούμενες αποδόσεις όσον αφορά ορισμένους τίτλους. Κυρίως μετά από την ε, περίπτωση που προσπαθήσαμε να αποφύγουμε, όπως γνωρίζετε, του PSI. για να χρησιμοποιήσω την σύντμηση που χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα στα αγγλικά. Το PSI λοιπόν με το οποίο οι αγορές θεώρησαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, είχε ένα καθεστώς ε, ε, προτιμούμενου πιστωτή, preferred creditor. Δεν συνέβη αυτό όπως γνωρίζετε, αλλά έτσι το ερμηνεύσαν οι αγορές και αυτό είχε συνέπειες σε αυτό το πρόγραμμα ειδικότερα. από τεχνική άποψη, θα το πω στα αγγλικά γιατί δεν γνωρίζω την ε, διατύπωση στα γαλλικά, υπάρχει το πρόβλημα του negative leverage, αρνητική μόχλευση που παρουσιάζεται σε αυτή την περίπτωση αγορά ενό συγκεκριμένου τίτλου από φορείς που εάν υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον δεν θα συμμετέχουν στο κόστος. Όλοι αυτοί λοιπόν οι προβληματισμοί είναι σημαντικοί για τη λήψη αποφάσεων που θα μπορέσουν ενδεχομένως να ληφθούν στο μέλλον ή όχι και τους σχετικούς συμβιβασμούς. Απλά ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην τεχνική πτυχή που είναι σημαντική. Θα ήθελα να αναφέρω για άλλη μια φορά ότι εμείς αυξήσαμε τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος μόνο κατά 500 δισεκατομμύρια και όχι κατά ένα τρισεκατομμύριο όπως ακούμε από ορισμένους κύκλους ναι, ένα τρισεκατομμύριο είναι το σύνολο δύο μακροπρόθεσμων ε, ε, πράξεων αλλά αυτό έγινε με μείωση άλλων ε, παροχών. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την εντολή μας, πρωταρχικός στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών. Σήμερα παρατηρείται ε, πληθωρισμός άνω του 2%. Κυρίως οι τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας γενικότερα Αναμένεται ότι από τις τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες το πετρέλαιο δεν θα συνεχίσει να αυξάνεται. Προβλέπουμε λοιπόν μείωση του πληθωρισμού ώστε από το πρώτο τμήμα του 2013 ο πληθωρισμός να έχει φτάσει κάτω από το 2%. Σήμερα όμως είναι πιο υψηλός Όταν παρατηρούμε τον πληθωρισμό αποκλείοντας τις τιμές των τροφίμων και της ενέργεια, το ποσοστό του πληθωρισμού ουσιαστικά είναι 1,5% αν δεν λάβουμε υπόψη τις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων. Πρόσφατα επαναλάβαμε πολλές φορές ότι βλέπουμε τώρα κινδύνους πληθωριστικούς ε, σχετικά ισορροπημένους. Ωστόσο, βλέπουμε και το έχουμε πει σαφώς κινδύνους για την ανάπτυξη. και πιθανή μείωση λόγω κινδύνων της ανάπτυξης. Δεν έχουμε πάψει να εξαρτώμαστε από το τι θα συμβεί στην οικονομία. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. εάν οι κίνδυνοι που έχουμε προσδιορίσει και αναφέρει υλοποιηθούν, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα προσαρμόσουμε την πολιτική μας όπως κάναμε και πέρυσι. Αυτό που συνέβη πέρυσι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, θα έλεγα, ...αυτής της αρχής ε, και της εφαρμογής αυτής της αρχής στο πρώτο μέρος του έτους... Ε, είχαμε μια οικονομική ανάκαμψη πληθωριστικοί κίνδυνοι υπήρχαν, αυξάνονταν και όλοι πίστευαν ότι η ανάπτυξη θα συνέχιζε διεθνώς. Όλος ο κόσμος αυτό πίστευε. Αρχίσαμε σιγά σιγά να τυποποιούμε να, την νομισματική μας πολιτική. Από τον Ιούλιο όμως και μετά και σε μεγάλο βαθμό λόγω του PSI για την Ελλάδα και διάφορα άλλα θέματα η κατάσταση αντιστράφηκε. Πρώτα στην Ευρώπη και στη συνέχεια σε διεθνές επίπεδο. Αμέσως εμείς προσαρμόσαμε την πολιτική μας. Πρώτα απ' όλα αυξήσαμε τα επιτόκια και μετά τα μειώσαμε. Αυτό αποδεικνύει ότι προσέχουμε διαρκώς τις εξελίξεις, ε, τις οικονομικές στο πλαίσιο της εντολής μας ε, και στο πλαίσιο των προοπτικών και της πολιτικής μας και προσαρμόζουμε έτσι την πολιτική μας. Μάλιστα, ας περάσουμε στο τέλος της συνεδρίασης. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνστάνσιο που παρευρέθηκε εδώ και μας εξήγησε την έκθεση και απάντησε τις διάφορες ερωτήσεις. Ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η έκθεση Ιδίας Πρωτοβουλίας για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα δώσουμε λεπτομέρειες αργότερα για τον ορισμό εισηγητών σκιωδών. Δεν έχουμε ακόμα λάβει κάποιες λεπτομέρειες πληροφορίες, αλλά θα ανακοινωθούν αργότερα. Διακόπτουμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε στις 3 η ώρα σήμερα το απόγευμα.